όλους τους συναδέλφους και πραγματικά συνεργάστηκα με αριθμούς συνεργάτες και άκουσα τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις τους ε, και η ομάδα της Επιτροπής Γεωργίας ε, αρίστευσε ως προς τις ικανότητες συνεργασίας και συντονισμού. Ευχαριστώ την Ανακαμίου, την προσωπική βοηθό μου, τη Γραμματεία της Επιτροπής Γεωργίας και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όχι μόνο τον Γενικό Διευθυντή αλλά και το επιτελείο του διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν διαθέσιμη, μας ε, προσκόμισε τα απαιτούμενα στοιχεία για να συντάξω την έκθεσή μου. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η εργασία αυτή είναι το προϊόν ε, ε, πολύμινης εργασίας, όπου όπως σας είπα ε, κάναμε δεκάδες συσκέψεις, συναντηθήκαμε με περιβαλλοντικές οργανώσεις, με συνεταιρισμούς γεωργών, γεωργών μη κυβερνητικέ οργανώσεις, μετήχαμε σε συσκέψεις, σε σεμινάρια, σε διάφορα κράτη-μέλη και γι' αυτό το λόγο αυτή η έκθεση απηχεί πέρα από την προσωπική μου άποψη αυτό που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την εξέβρεση μιας πολιτικής ε, συμβαστικής ε, λύσης. Αν φυσικά δεν είχα άλλους περιορισμούς ε, και συνέτασα την έκθεση μου Εκφράζοντα μόνο τη δική μου άποψη θα ήταν τα πράγματα διαφορετικά αλλά ε, πιστεύω ότι αυτή η έκθεση που είναι προϊόν ε, αυτή τη συνεργασία ε, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για το μέλλον αποτυπώνει την αρχιτεκτονική που εισηγήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο σύστημα και ταυτόχρονα προσπαθούμε να προωθήσουμε μια, ένα πιο ρεαλιστικό μοντέλο για να επιτύχουμε του ίδιου στόχου, δηλαδή να είναι πιο δίκαιη η νέα κοινή γεωρική πολιτική και κυρίω να είναι απλούστερη η εφαρμογή να μειώσουμε την γραφειοκρατία και να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή ανάμεσα στους δύο πυλώνες ε, της κοινή γεωργικής πολιτικής. Και γι' αυτό έφερα αυτήν την διητή ευθύνη ως εισηγητής ε, και υπάρχουν ε, πάρα πολλές διασυνδέσεις ανάμεσα στους δύο πυλών. Σας αρχίσω με τον πρώτο. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομο γίνεται, αλλά θα ήθελα να εξηγήσω τα βασικά στοιχεία που εισηγούμε. Λοιπόν, ο ενεργό γεωργό είναι μία έννοια που είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη. Ήταν ιδιαίτερα δυσχερή η εξέβρεση μια συμβαστική δυσχερής η εξεβρεση μια συμβαστικη λυση σε ευρωπαϊκή κλίμακα, δοθέντω του ότι Κάποια κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύουν ότι ο ενεργός γεωργός θα πρέπει να οριστεί με διαφορετικό τρόπο από αυτό που προτιμούν κάποια άλλα κράτη-μέλη. Δηλαδή, ο ενεργός γεωργός ποιος είναι. Αυτός που έχει την γεωργική δραστηριότητα ε, ως βασική του δραστηριότητα, όταν δηλαδή ε, απασχολείται και σε άλλους τομείς, το καθεστώς αυτό σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσδιοριστεί σε επίπεδο κράτους μέλους επί τη βάση αυτής της γενικής αρχής, δηλαδή ότι ο ενεργός γεωργός είναι ο γεωργός που έχει γεωργική δραστηριότητα και είναι η βασικότερη των δραστηριοτήτων τους. Στη συνέχεια, ως προς τον αρνητικό κατάλογο σχετικά με τις ε, γέ τα αγροτεμάχια που δεν θα είναι επιλέξιμα για τις άμεσες πληρωμές, ε, διότι πρόκειται για εδάφη που καλλιεργούν για κάποιους άλλους λόγους. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα, ε, αθλητικές δραστηριότητες, ε, ορυχεία, αεροδρόμια, όλα αυτά τα αγροτεμάχια που μέχρι στιγμής ήταν επιλέξιμα για την επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα πρέπει να αποκλειστούν. Ένα άλλο επίσης αφιλεγόμενο ζήτημα είναι τα ανώτατα όρια και ε, η φθήνουσα πορεία των πληρωμών. Εν μέρη προσυπογράφουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όμως στην έκθεσή μας προτείνουμε κάποιες διορθώσεις που είναι δικαιότερες ε, κατά τη γνώμη μας. Παραδείγματος χάρη, προσδιορίζεται με σαφήνεια ότι η μείωση των ποσών είναι εφαρμοστέα σε κάθε, ε, σε κάθε μία από τις κλίμακες πάνω από τις 150.000 ευρώ. Όταν μιλάμε για το μείον 20% των επιδοτήσεων, ε, λοιπόν ε, μιλάμε για ένα ποσό που τοποθετείται στην ψαλίδα από 150.000 μέχρι 200.000 ευρώ και όχι κάτω των 150.000 ευρώ. Συνέχεια έχουμε το ανώτατο όριο των 300.000 ευρώ είναι ένα μέτρο που εξασφαλίζει μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Θεωρώ ότι αυτό το ανώτατο όριο είναι υψηλότερο σε σχέση με το αμερικανικό σύστημα όπου υπάρχει ε, ένα αντίστοιχο όριο που κυμαίνεται στις 250.000 δολάρια. Τώρα, σε σχέση με την ευελιξία για τη διασύνδεση των δύο πυλώνων, πράγμα που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη γνώμη μου, Λοιπόν, προτείνω το εξή. Τα κράτη-μέλη που έχουν περιέλθει σε μια δυσμενέστερη θέση ε, στο εσωτερικό του ε, δεύτερου πυλώνα είναι τα κράτη-μέλη που βρίσκονται σε ευμενέστερη θέση στον πρώτο πυλόν. Οπότε εγώ προτείνω οι μεταφορές ε, ανάμεσα στους δύο πυλώνες, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, αυτά είναι τα 7 κράτη-μέλη, μπορούν λοιπόν να μεταφέρουν από τον ένα πυλώνα στον άλλον μέχρι 20%. Ο πρώτος πυλώνας λοιπόν είναι άνετο, σας το εκφράσω έτσι, και θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν μεγαλύτερες πιστώσεις στο δεύτερο πυλώνα, ώστε να ε, περατωθεί επιτυχώς η πολιτική ανάπτυξη υπαίθρου αυτών των κρατών. Στη συνέχεια τα κονδύλια του πρώτου πυλώνα που δεν χρησιμοποιούνται και προορίζονται στις ε, περιοχές που βρίσκονται στη δυσμενέστερη θέση θα πρέπει να μεταφέρονται στο δεύτερο πυλώνα, δηλαδή ότι δεν χρησιμοποιείται για το πρασίνισμα του πρώτου πυλώνα θα πρέπει να μεταφέρεται στο δεύτερο πυλώνα για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Τώρα σε σχέση με το καθεστώς της βασικής πληρωμής που ενδέχεται να ενεργοποιηθεί για κάποιους γεωργούς όταν ενεργοποιούνται αυτά τα δικαιώματα δεν θέλουμε να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο σύγκρισης μόνο το 2011 ε, θα πρέπει να δοθούν οι λόγοι για τους οποίους δεν ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός το 2009 και το 2010 ούτω ώστε να αποδειχθεί η βασική δραστηριότητα αυτών των γεωργών. Κάτι άλλο τώρα που επίσης είναι αφιλεγόμενο είναι το πρασίνισμα, αυτό καθεαυτό. Όλοι μας θέλουμε να είναι πρασινότερη η κοινή γεωργική πολιτική στον πρώτο πυλώνα και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Όμως, οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, αφενός ε, αποδεικνύονται δυσεφάρμοστες ε, και είμαι πεπισμένος ότι συνεπάγονται ένα μεγαλύτερο γραφειοκρατικό άχθος. Αφήστε που ήταν η τα μέτρα της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, εγώ εισηγούμε νέα μέτρα και διόρθωση υφιστάμενων μέτρων. Ως προς τα νέα μέτρα που προτείνω, προτείνω το εξή. Ε, επιλεξιμότητα ύψο φάκτο των ε, επιφανειών που είναι επιλέξιμες για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα του τέστην. Τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα ε, θα εξυπηρετούν τον ίδιο στόχο που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Βιολογική Γεωργία. Στο δεύτερο πυλώνα, στην ανάπτυξη δηλαδή της υπαίθρου, τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα υποχρεωτικά θα πρέπει να έχουν μια ακόμη πρασινότερη διάσταση σε σχέση με τον πρώτο πυλώνα. Αυτή η υποχρέωση ε, διευκολύνει του γεωργού και καθιστά ακόμη πιο υποχρεωτικό το πρασίνισμα του δεύτερου πυλώνα. Στη συνέχεια, ένα ρηξικέλευθο μέτρο προτείνω την οικολογική πιστοποίηση με ισοδυναμία ως προς το πρασίνισμα. Τι εννοώ. Με το που προσδιορίσουμε ένα ευρωπαϊκό ενίο πλαίσιο που επιτρέπει ότι κάθε κράτος μέλος μπορεί να προβεί σε οικολογική πιστοποίηση των καλλιεργειών, αυτό μας επιτρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες σε κάθε περιοχή και κάθε κράτος στο πλαίσιο του πρασινίσματος συμπληρωματικά σε σχέση με τα μέτρα που μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο μέτρο που αυτό το μοντέλο πιστοποίησης θα πλαισιώνεται και το τονίζω αυτό ε, από ευρωπαϊκές διατάξεις. Ε, άλλο νέο στοιχείο, η δυνατότητα επιλεξιμότητας ε, για άμεσους πληρωμές, δηλαδή πρασίνισμα των μονίμων καλλιεργειών, όχι μόνο τα μόνιμα σκοτόπια αλλά και τις μόνιμες καλλιέργειες όπως το αμπέλι, οι ελιές, τα απορροκυπευτικά ε, και εδώ έχουμε μια διάσταση προστασίας ε, του εδάφους και γι' αυτό σας λέω ότι τονίζεται το, η πτυχή του πρασινίσματος. Επίσης, Προτείνω απλούστευση αρκετά μεγάλη των ε, μέτρων παρασυνίσματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ας αρχίσουμε τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών, την σπόρα Μέχρι, τις 5, μέχρι τα 5 εκτάρια προτείνω να μην απαιτείται από τους γεωργούς να εφαρμόζουν αυτά τα μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την εξαίρεση μόνο ε, για... Ε, Επιφάνει κάτω των 13 εκταρίων. Εγώ προτείνω αλλαγή του ορίου στα 5 και προτείνω στα στις ε, επιφάνειες από τα 5 έως τα 20 εκτάρια να είναι υποχρεωτικές σε δύο διαφορετικές καλλιέργειες και όχι τρεις. Ε, ε, σε επιφάνειες κάτω των 5 εκταρίων δεν θα υπάρχει η υποχρέωση των δύο καλλιεργειών όταν το 80% της αρρώσιμης γης καλύπτεται από μόνιμες καλλιέργειες. Αυτό το μέτρο, κατά τη γνώμη μου, απλουστεύει πάρα πολύ το σύστημα διότι μιλάμε για το 80% τη της αλλά δεν αποκλείουμε το 80% των γεωργών, αποκλείουμε το 20% μόνο τη έκταση. Ε, άρα ε, το πρασίνισμα ενισχύεται, διότι καλύπτουμε το 80% τη καλλιεργήσιμης γης Ευρωπαϊκής Ένωση, ε, ανερώντας όμως και καταργώντας όλη τη γραφειοκρατία που φέρουν στους ώμου τους οι γεωργοί. Σε σχέση τώρα με τις μόνιμες καλλιέργειε, προτείνουμε ε, με ένα σύστημα που προσωμιάζει αυτόν τον βόσκο Τι εννοώ. Ε, υπάρχει ε, η έννοια του ε, μόνιμου βοσκοτοπιού που καλύπτει περιοχές όπως παραδείγματος χάρη η Βάλτη της Σκοτίας. τώρα ε, οι περιοχές οικολογικής εστίασης. Εγώ προτείνω να παραμείνει το 7% για την καλλιέργεια που μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά στη συνέχεια θέλω να εφαρμόζεται αυτό ε, σε επιφάνεια άνω των 20 εκταρίων. Και πάλι εδώ ο στόχος ε, δεν είναι να αποκλείσουμε το 80% των γεωργών, αλλά να αποκλείσουμε μόνο το 20% της καλλιεργήσιμης μυσηγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η περιοχή περιοχή οικολογικής εστίασης μπορεί να αντικατασταθεί από καλλιέργειες που δεσμεύουν τα οξύδια του αζότου. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε αυτές τις καλλιέργειες προστατεύοντας το έδαφος ε, και ο βασικός λόγος είναι ότι έτσι ε, καταπολεμούμε και το έλλειμμα σε πρωτεΐνες ε, που πλήττει την Ευρωπαϊκή Ένωση, φυτικές πρωτεΐνες. Κάθε φορά λοιπόν που ε, οι γεωργοί έχουν ε, δύο τέτοιες ε, καλλιεργήσιμες ε, εκτάσεις, τότε θα ισχύει το όριο του 5% για να συνδυαστούν και να υπαρθούν στο ίδιο καθεστώς οι δύο καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Ως προς τους νέους γεωργούς, προτείνω να διατηρηθεί το 25% της προσάυξησης της άμεσης πληρωμής, ακριβώς όπως το προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως η προσάυξηση αυτή θέλουμε εμείς να περιοριστεί στα 50 εκτάρια για όλους τους Ευρωπαίους γεωργούς και όχι να προσαρμόζεται ε, και να υπολογίζεται η αξία της βάσει του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας γεωργός, οποιοδήποτε κράτους μέλος, πλήττεται σε σχέση με κάποιον άλλον και βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση, διότι ο μέσος όρος της ε, καλλιεργήσιμης έκτασης ε, στη χώρα του άλλου γεωργού είναι ανώτερη. Οπότε έχω προτείνω για τους νέους γεωργούς να διατηρηθεί το ίδιο ποσοστό του 5%. Στη συνέχεια προτείνω η εισαγωγή του συντελεστή της εργασίας ε, ως μία από τις προϋποθέσεις ε, βάση των οποίων το κράτος ε, κρίνει αν θα χορηγήσει τις άμεσες πληρωμές επί τη βάση της παραγωγής. Δηλαδή υπάρχουν οικονομικοί λόγοι, υπάρχουν ε, παραδείγματο χάρη λόγοι που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο οικονομικό τομέα, οπότε το κράτος μπορεί να αποφασίσει για μία περιοχή ότι ο συντελεστής εργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός και εισάγοντας αυτόν τον νέο συντελεστή κάθε κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα της συνδεδεμένη πληρωμής φυσικά μέσα στα ε, διορισμένα εκ των προτέρων σωστά. Στη συνέχεια, οι γεωργοί θα μπορέσουν με τα μέτρα μας ε, ε, να αναβαθμιστούν ως προς την ποιότητα ζωή τους, ε, διότι προτείνουμε τα 1500 εκτάρια παραδείγματο χαρή για του νέου μικρού γεωργού. Αλλά θέλω να διευκρινίσω εδώ ότι τα κράτη-μέλη δεν συμφωνούν επ' αυτού και θα Ήθελα να εισηγηθώ να έχει προαιρετικό χαρακτήρα αυτό το μέτρο, όχι υποχρεωτικό όπως ε, ε, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, είναι μια πολιτική συμβαστική λύση γιατί αν διατηρήσουμε υποχρεωτικό το σύστημα θα έχουμε ζήτημα σε σχέση με τα ανώτατα όρια. Δηλαδή υπάρχουν κράτη-μέλη που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο αλλά αφήνουμε ταυτόχρονα την ελευθερία σε άλλα κράτη-μέλη να μην ακολουθήσουν αυτό το δρόμο αν δεν το κρίνουν απαραίτητο. το πλέον πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα, δηλαδή τα ανώτατα εθνικά όρια και ανακατανομή των κονδυλίων, εγώ προτείνω ένα μηχανισμό που μου φαίνεται δικαιότερο σε σχέση με αυτόν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζουμε όλοι ότι η κοινή γεωργική πολιτική είναι άδικη για πολλά κράτη-μέλη και για πολλέ περιοχέ. Για ιστορικού λόγου υφίστανται ακόμη πελώριε διαφορέ ω προ τη μέση πληρωμή ανά εκτάριο και γνωρίζουμε ότι από πολιτική σκοπιά ε, θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια ρότα που θα ε, αμβλύνει αυτές τις ε, μεγάλες διαφορές. Οπότε ε, θέλουμε να καταπολεμήσουμε την αδικία αυτή ε, εις βάρος σε κάποιων κρατών μελών. Υπάρχουν ακραίες όμως περιπτώσεις. Κάποια κράτη-μέλη λαμβάνουν πάνω από 60% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα κράτη-μέλη που λαμβάνουν το ίμιση e του μέσου όρου ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι φυσιολογική αυτή η κατάσταση. Προτείνω λοιπόν στα κράτη-μέλη, τα κράτη-μέλη που βρίσκονται στη δεσμενέστερη θέση και οι σε χώρες είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα να μπορέσουν να υποφεληθούν από το νέο καθεστώ και να κάνουν περισσότερε θυσίε. στα κράτη-μέλη που βρίσκονται πάνω από τον μέσο όρο, τον ευρωπαϊκό, βάσει του εθνικού κονδυλίου που έχουν. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν στον πρώτο πυλόν ένα μεγαλύτερο ε, ποσοστό ε, των επιδοτήσεων. Αυτά τα κράτη-μέλη λοιπόν που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό θα πρέπει να θυσιαστούν ούτω ώστε να καλυφθεί αυτό το έλλειμμα, αυτό το χάσμα με τα κράτη-μέλη που βρίσκονται κάτω από το 70% ε, ε, του κοινοτικού μέσου όρου. Δηλαδή μέχρι το 2019 θα πρέπει να ανέβουν αυτά τα κράτη-μέλη κατά 30% σε σχέση με την τωρινή τους ε, κατάσταση. Άρα σύγκληση προς τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι σύγκληση προς το 90% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα κράτη-μέλη που βρίσκονται ανάμεσα στο 70% και 80% του μέσου μέσου όρου ε, θα ε, προτείνουμε να ε, αυξηθεί αυξηθούν κατά 25% και όσα κράτη-μέλη βρίσκονται ανάμεσα στο 80% και ε, το 100% θα μπορούν ε, να αυξήσουν τις επιδοτήσεις μόνο κατά 10%. Ε, αφετέρου, ω προς τη σύγκληση των πληρωμών στο εσωτερικό του ίδιου κράτου μέλους, όπερ και είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα για κάποια κράτη όπου υπάρχουν τομείς, όπως παραδείγματο χάρη ιδιαίτερα διαφοροποιημένη γεωργία ή τομείς όπου οι πληρωμές είναι ιδιαίτερα υψηλές, όπως γαλακτοκομικός τομέα για κάποια κράτη-μέλη. Λοιπόν, προτείνω άμεση μείωση σε σχέση με αυτό που μα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περικοπέ ε, δηλαδή σε κάποιους τομείς ε, και σε κάποια ε, κράτη-μέλη για να διορθωθεί η κατάσταση προτείνω έναν αναλλακτικό μηχανισμό που μπορούν να ενεργοποιήσουν αυτά τα κράτη-μέλη που έχουν τις μεγαλύτερες, τα μεγαλύτερα προβλήματα. Δηλαδή να θέσουν ένα ανώτατο όριο το 30% μέχρι το 2019 για τις άμεσες πληρωμές. Δηλαδή τα κράτη-μέλη θα ξέρουν ποιο είναι το ανώτατο όριο της περικοπής των βασικών τους πληρωμών για την ε, περίοδο αυτή μέχρι το 2019 και πάλι επιδιώκονται σύγκληση ανάμεσα στα κράτη-μέλη επιταχύνονται τη διαδικασία σε σχέση με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προτείνω και σύγκληση στο εσωτερικό του κράτου μέλους με μικρότερη όμω ταχύτητα σε σχέση με αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, δεν είναι λογικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδιώκει τόσο μεγάλη σύγκληση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα στο εσωτερικό των κρατών μελών, ενώ ταυτόχρονα είναι βραδύτατη η προσαρμογή και η σύγκληση που προτείνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και γι' αυτό ε, αυξομειώνουμε την ταχύτητα ανάλογα με το αν μιλάμε για το ιστορικό του κράτους μέλους ε, ή για, τις, ε, για το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για όλα τα κράτη-μέλη, για να καταστεί δικαιότερο το σύστημα. Προτείνω λοιπόν αυτές τις αλλαγές για τον κανονισμό που διέπει τις βάσικες πληρωμές. Τώρα θα εντάχει, ας περάσω και στην ανάπτυξη της υπαίθρου, διότι υπάρχουν κάποιες διαστάσεις του ζητήματος που συνδέονται και με τον κανονισμό των άμεσων πληρωμών. Αρχίζω λοιπόν από τους νέους γεωργούς οι νέοι γεωργοί, όπως ε, λέγαμε και για τον πρώτο πυλώνα, ε, θα πρέπει να έχουν την προσάυξηση, το top-up, το 25% μέχρι τα 50 εκτάρια για όλα τα κράτη-μέλη. Στο δεύτερο πυλώνα, ως νέο στοιχείο, προτείνω να καταστούν επιλέξιμες πληρωμές που σχετίζονται με τις προσόδους ε, της γης. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα του νέου γεωργού είναι η πρόσβαση στα αγροτεχνικά τεμάχια τα οποία είναι ιδιαίτερα ακριβά, δεν είναι ε, πάρα πολύ εύκολο να αρχίσει κανείς ε, να ασκεί αυτό το επάγγελμα δεν έχει κληρονομήσει παραδείγματος χάρη τα αγροτεμάχια από την, ε, από την οικογένειά του. Έτσι διευκολύνουμε την πρόσβαση των νέων γεωργών στην υγεία και ταυτόχρονα εισάγουμε νέο μηχανισμό παύσης της δραστηριότητας. Πρόκειται για μία απλή μεταρρύθμιση που είναι ευεφάρμοστη. Προτείνω λοιπόν οι γεωργοί που είναι πάνω από 65 ετών να λαμβάνουν μία ενιαία πληρωμή που αντιστοιχεί στο 50% της επιδότησης εγκατάστασης του νέου γεωργού εάν μεταβιβάσουν την έκταση και τα δικαιώματα πληρωμής είτε στο νέο γεωργό είτε σε ένα σε έναν άλλο γεωργό με αυτό το σύστημα που προτείνουμε ανανεώνεται ο πληθυσμός των γεωργών. Ε, αφετέρου, ε, θέλουμε να διευκολύνουμε την αναδιάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ε, προτείνοντας μία εφάπαξ πληρωμή που αντιστοιχεί στο ποσό της πενταετίας για τους νέους γεωργούς που αποφασίζουν να πάψουν τη δραστηριότητά τους προσαυξάνοντας κατά 20% την ενιαία πληρωμή. Δεν θέλω τώρα να πω σε τεχνικά ζητήματα, αλλά ουσιαστικά περί πρόκειται μία εφάπαξ πληρωμή για ένα νέο γεωργό προσαξιμένη κατά 20% στο μέτρο που ε, γίνεται μεταβίβαση της καλλιεργούμενης έκτασης ή των δικαιωμάτων πληρωμής. Στη συνέχεια διευρύνω την επιλεξιμότητα ως προς τις επενδύσεις που γίνονται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στην αγροβιομηχανία. Θεωρώ ότι ε, επιβάλλεται αυτό στο μέτρο που υπάρχει μια νέα αγροπεριβαλλοντική ε, ή φυτογειονομική απέτηση βάσει του νέου κανονισμού. Εν τη αυτή περιπτώσει στην πολιτική ανάπτυξη υπαίθρου θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για επιδότηση οι καλλιεργούμενε εκτάσει. Είχα, ε, είχα προτείνει συγγνώμη, την, τον αποκλεισμό των παλιών κρατών μελών ω προς επιδοτήσει για τι επενδύσει και τι νέε αρρώσιμες γέε. κυρίως ε, για τα κράτη-μέλη του Νότου, όπου δύσκολα μπορεί να γίνει ανταγωνιστική η γεωργία χωρίς ε, την κατάλληλη άρδευση. πιστεύω ότι θα πληγούν ιδιαίτερα αυτά τα κράτη-μέλη και ως εκ τούτου θεωρώ ότι η επιλεξιμότητα για τις νέες επενδύσεις ε, θα πρέπει να εξακολουθήσει να υπάρχει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλο ένα νέο στοιχείο για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα είναι το εξής, τουλάχιστον 30% ε, του προϋπολογισμού της ανάπτυξης υπαίθρου θα έπρεπε κατά τη γνώμη μα να συνδεθεί με αυτά τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λογικό διότι όταν συμπεριλαμβάνουμε τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα στο πρασίνισμα είναι απαραίτητο στο δεύτερο πυλώνα να έχουμε και τα απαιτούμενα κονδύλια, την απαιτούμενη χρηματοδότηση. Τα κράτη-μέλη τουλάχιστον 30% πρέπει να αφιερώσουν σε αυτό τουλάχιστον το 1 τρίτο δηλαδή του γενικού κονδυλίου θα πρέπει να διοχετεύεται σε αυτά τα μέτρα, γιατί από οικολογική σκοπιά ε, θα είμαστε έτσι πιο απαιτητικοί σε σχέση με οποιοδήποτε μέτρο πρασινίσματος ε, εισάγουμε στον πρώτο πληρών ε, επίσης προτείνουμε ε, το φάσμα των επιδοτήσεων να καλύπτει και την δασοκομεία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας προτείνει άλλες κατηγορίες γεωργών όπως παραδείγματος χάρη ε, τα κοινά δασίλεια, ε, ε, ούτε τα ιδιωτικά ούτε τα δημόσια να μπορέσουν να ενταχθούν παραδείγματος χάρη σε αυτό το σύστημα. Μία άλλη, θα το πω, πιο επαναστατική ιδέα ή πιο αμφιλεγόμενη, όπως θέλετε πείτε το, σε σχέση με την ανάπτυξη της υπαίθρου σχετίζεται με τις ζώνες που υπάγονται σε ιδιαίτερους ε, περιβαλλοντικούς ε, όρους. Ε, είναι ιδιαίτερα λεπτό το ζήτημα, διότι πάνω από 10 κράτη-μέλη δεν κατέφεραν μέχρι του δεν να αναλύσουν τις άμεσες επιπτώσεις εφαρμογής των κριτηρίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον γεωγραφικό προσδιορισμό των ζωνών αυτών. Δεν φαίνεται δίκαιο ούτε και ηθικά αποδεκτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δίνεται να αποφασίσει για, μη, ένα μέτρο ε, του οποίου τις επιπτώσεις αγνοεί. Και γι' αυτό σας προτείνω ε, να λάβουμε υπόψη την ομολογία ε, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Αυτές οι ζώνες ε, λοιπόν με ιδιαίτερους οικολογικούς όρους πρέπει να προσδιοριστούν επί τη βάση βιοφυσικών κριτηρίων αποκλειστικά και μόνο χρησιμοποιώντας τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως δείκτες και όχι ως υποχρεωτικά κριτήρια. Αυτή είναι η δική μας πρόταση, ώστε να έχουν μεγαλύτερο περιθώριο, ε, μεγαλύτερη ευχέρεια να κινηθούν και μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών τα κράτη-μέλη σε σχέση και με τις απαιτήσει ε, του ΠΟΕ. Ε, για την διαχείριση των κινδύνων τώρα υποστηρίζω την Ευρωπαϊκή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ταυτόχρονα όμως ε, μιλώ για τα ταμεία άλλη ούτως ώστε ε, να αντιμετωπίσουμε ε, ένα φαινόμενο που πλήττει τις νότιες χώρες με κυκλικό τρόπο, δηλαδή οι ξηρασίες και όχι μόνο όποια θεωρούμε ότι αυτά τα ταμεία αλληλασφάλισης μπορούν να μας βοηθήσουν να ενταχθούν στο σύστημα ε, διαχείρισης ετών και να αντιμετωπίσουμε αυτό το ιδιαίτερο φαινόμενο. Τώρα, συντελεστή σε συγχρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτείνει 60% ε, και 80% από 50% σε 60% και από 85% σε 90% ε, για αφενός ε, ε, το μέσο όρο των κοινοτικών και αφετέρου τις εξαιρετικά απομακρυσμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρα από τις αλλαγές των ποσοστών προτείνω ό,τι δεν χρησιμοποιείται στο πρασίνισμα του πρώτου πυλώνα να μπορεί να μεταφερθεί στο δεύτερο πυλώνα. Σε σχέση τώρα με τον προϋπολογισμό αυτών καθεαυτών της ανάπτυξης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε προτείνει συγκεκριμένο προπολογισμό και εμεί επικρίνουμε το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει συγκεκριμένο ε, προπολογισμό για τον πρώτο πυλώνα, αλλά όχι για τον δεύτερο. Ε, αναέλυσα ε, διάφορα εναλλακτικά σενάρια και κάναμε επί χάρτου διάφορε ασκήσει ανακατανομή των κονδυλίων. Λοιπόν, ε, στο δεύτερο πυλώνα, τα κράτη-μέλη που βρίσκονται στην ευμενέστερη θέση στο δεύτερο πυλώνα είναι, αυτές που βρίσκονται, είναι αυτά που βρίσκονται σε ευμενέστερη θέση στον πρώτο πυλώνα. Τι γίνεται. Ε, στις βαλτικές χώρες, στην Πολωνία, στη Ρουμανία. Ε, βάσει αυτού του σύμφωνο που μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι δυνατή η μεταφορά πιστώσεων προς χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία ε, προσπαθούμε να εξισώσουμε τη θέση των κρατών μελών και πιστεύω ότι ανακατανέμοντας ένα μικρό κομμάτι των κονδυλίων των μεγάλων κρατών μελών που όντω βρίσκονται στη χειρότερη θέση στο δεύτερο πυλώνα μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα κονδύλια των κρατών μελών που βρίσκονται στην καλύτερη θέση στον πρώτο πυλώνα και προτείνω νέα κλίδα ανακατανομής συμπληρωματική ως προς ε, την υφιστάμενη διότι ε, δεν συντρέχουν λόγοι ούτως ώστε να προτείνω ουσιαστικά ουσιαστική ε, τροποποίηση της φυστάμενης κλίδας ανακατανομής. Ε, αυτές είναι οι βασικές μου προτάσεις, ε, Πρόεδρε. Αναμένω την δική σας συμβολή. Όπως και μέχρι στιγμής θα σας ακούσω με προσοχή, διότι συνεχίζει η διαδικασία διαπραγμάτευσης και οποιαδήποτε δικό σας σχόλιο θα εμπλουτίσει την συζήτηση και σας ευχαριστώ και πάλι κλείνοντας για τη συνεργασία σας μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ. Bene, grazie Luis, hai fatto davvero un lavoro importante. Eh, Πολύ σημαντική η δουλειά σου, Λουίς. Ελπίζω ότι η ενσωμάτωση πολλών γνωμοδοτήσεων μέσα στην έκθεσή σου θα βοηθήσει ιδιαίτερα αυτή η ένταξη για τις συζητήσεις. Θα κάνουμε ό,τι κάναμε και χθε με τον Μισελ Νταντέν και με τον ε, Λαβία. Οπότε θα γίνει συζήτηση. Ξεκινάμε με τις άμεσες ε, βοήθειες. Η Μάριον Μαγκίνες και μετά ο Τζορτζ Λάιον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή για την ε, παρουσίασή του, τη σαφήνεια, αλλά βέβαια και τη μέθοδο εργασίας του. Οπωσδήποτε μας άκουσε όλους και έλαβε υπόψη κάποιες ανησυχίες μας. Ευχαριστώ λοιπόν κύριε. Κύριε Πρόεδρε, πόση ώρα έχω. Ε, σκοπεύω να είμαι σύντομη. Σημαντική ερώτηση, λέει ο Πρόεδρος. Για τους οικειώδες χθες ε, δεν είχαμε χρόνο, οπότε... Και ούκαν το πολλό το εφ, ξέρετε. Θα προσπαθήσω να είμαι κάπως ε, σύντομη. Λοιπόν, να ξεκινήσω με κάποια ζητήματα. Για το πρασίνισμα, καλώς ορίζουμε κάποιες προσπάθειές σας για τους μικρότερους ε, αγρότες, αλλά πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες. Κάτι το οποίο θέλω να πω. Είχε ψηφίσει το Κοινοβούλιο ένα σύστημα μενού με κάποιες επιλογές πρασινίσματος για να διαλέγουν τα κράτη-μέλη ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους. Αυτό δεν είναι στην έκθεση, δεν ξέρω το εξετάσατε γιατί δεν είναι μέσα. Είναι κάτι το οποίο νομίζω θα θέλαμε να επανεισαχθεί για να έχουμε μέτρα πρασινίσματος τα οποία θα ταιριάζουν στο κάθε κράτος μέλος ε, για την ε, άμυψη σφορά ξέρουμε πως είναι καλύτερο μέτρο όσον αφορά την εναλλαγή των καλλιεργειών. Τώρα για τις ε, περιοχές οικολογικής εστίασης υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν σοβαρά προβλήματα. Οι συνάδελφοι από τη Γερμανία που ανησυχούν για το 7% αλλά η ιδέα ίσως είναι καλή. Γι' αυτό ίσως ε, το σύστημα αυτό του μενού που ανέφερα ε, μπορεί να κάνει αυτό το πρασίνισμα να λειτουργήσει. Όσον αφορά τις ιδέες τώρα. Νομίζω πως πάμε Συμβούλιο και Κοινοβούλιο και η Κομισιόν ε, προς ε, μια κατεύθυνση να βελτιώσουμε τα του πρασινίσματος, αλλά έχει, έχουμε πολύ δουλειά ακόμα να κάνουμε γιατί σας άκουσα να μιλάτε για όρια στρεματικά και ποσοστά. Καλό να ακούσουμε και τους αγρότες ε, εδώ μέσα και εκτός βεβαίως για να μας πούν πώς θα ε, προσαρμοστούν σε αυτές τις δύσκολες ε, συνταγές εδώ πέρα και πώς θα μπορούν να καλλιεργήσουν υπ' αυτές τις συνθήκες. Τα μέτρα αυτά λοιπόν δεν είναι απλοποίηση, κάνουν τα πράγματα πιο πολύπλοκα. Ένα τελευταίο σχόλιο για το πρασίνισμα και ο Λουίς το γνωρίζει αυτό. Υπάρχει σχέση μεταξύ πυλώνα 1 και 2. Πώς αποφεύγουμε το πρόβλημα των διπλών πληρωμών ενώ ταυτόχρονα αποδεχόμαστε ότι αυτομάτως συμπεριλαμβάνονται οι βιολογικές καλλιέργειες. Θέλουμε να συμπεριλάβουμε και όσου είναι στα αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα και υπάρχει και η πρότασή σας να συμπεριληφθεί και η πιστοποίηση. Νομίζω πως η Κομισιόν πρέπει να το δει αυτό το θεμελιώδες ζήτημα του πώς θα αποφύγουμε τις διπλές πληρωμές ή αν πρέπει να αποφευθούν οι διπλές πληρωμές. Και επιπλέον πώς θα διασφαλίσουμε πως ε, θα έχουμε σωστά συστήματα αγροτοπεριβαλλοντικά στον πυλώνα 2, ενώ θα υπάρχει και ο πυλώνα 1, γιατί όπως θα ξέρουν οι συνάδελφοι, το πρασίνισμα θα γίνει η βάση από ό,τι καταλαβαίνω των αγροτοπεριβαλλοντικών του πυλώνα 2 και αυτό είναι επικίνδυνο. Καλό είναι να μας πει κάτι ο εισηγητής και η Κομισιόν. Για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Δεύτερον, για τα σχόλια που έκανε ο Πρόεδρος για τον προϋπολογισμό. Ίσως από εκεί έπρεπε να έχουν ξεκινήσει. Θα ήμασταν πολύ δικαιότεροι εάν είχαμε ένα σωστό προϋπολογισμό. Και η ανησυχία μας εκφράστηκαν, ανησυχούμε για το ότι θα υπάρχουν λιγότερα χρήματα και βεβαίω βασιζόμαστε στον Πρόεδρό μας για να υπερασπίσει τον ρόλο του Κοινοβουλίου στον προπολογισμό. Αλλά ανησυχώ ιδιαίτερα. Οπότε, το ζήτημα της κατανομής μεταξύ κρατών μελών και εντός των κρατών μελών γίνεται πολιτικά ευαίσθητο και νομίζω πως εργάζεται προς μια κατεύθυνση για να αντιμετωπίσετε τις ανησυχίες ε, αυτών που έπαιρναν πάρα πολύ λίγα από τις άμεσες πληρωμές αλλά το κάνετε με λιγότερα λεφτά και νομίζω πως εδώ είναι η δυσκολία μας και θα υπάρχουν πολιτικά προβλήματα και στις 27 χώρες μας. Γιατί Μιλάμε για έναν προπολογισμό μειωμένο. Αλλά σας συγχαίρω για το ότι θέλετε να ξαναδείτε την ε, συνταγή, τον τύπο. Τώρα για να κατανοούμε μεταξύ κρατών Ξέρω πως θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μια ισοπαίδωση με τον τρόπο που προτείνει η Κομισιόν Νομίζω πως ε, εσείς αντιμετωπίζετε με τρόπο θετικό, αναγνωρίζετε με τρόπο θετικό το πρόβλημα. Για τις ε, πράσινες πληρωμές ε, ασχοληθήκατε ειδικά με τη βασική πληρωμή και προσπαθήσατε να μειώσετε, να αυξήσετε τον χρόνο αναδιανομής εσωτερικά, αλλά δεν έχετε λάβει υπόψη το τι θα σημάνει η πληρωμή αυτή κατά αποκοπήν θα ήθελα και εδώ πέρα κάποιο σχόλιο. Επίσης μπορούμε και εμείς ε, να δούμε κάποιες άλλες ε, μεθόδους για τις πράσινες ε, πληρωμές. Πρέπει να είναι μια πληρωμή κατά σε όλες τις εκτάσεις. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε και ξέρω πως δεν συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι να επιτρέψουν σε όλα τα κράτη-μέλη που έχουν κάποια ιστορία να έχουν μακρύτερη περίοδο για να διανομή. Θα μπορούσαμε να βρούμε κάποιο βασμό, αλλά συνοψίζοντα όπω είπα, υπάρχουν 27 χώρε. ως 27 άλογα, σαν να ήταν 27 άλογα, αν θέλετε, που ξεκινάνε όμω τον αγώνα από διαφορετικά σημεία τη ε, ε πίστα του υποδρομίου. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς ε, θα καταφέρουμε να τερματίσουμε. Αλλά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε εντό χρόνου διαγράμματος του Τελικομισιόν. Κάποια άλλα πράγματα για την ε, στήριξη, την συνδεδεμένη. Μιλήσατε για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής. Ε, υπάρχει οπωσδήποτε στις περιφέρειες κάποιος ρόλος που έχει να παίξει η συνδεδεμένη ε, ενίσχυση Επίσης σας στηρίζω για τους νέους αγρότες, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την εφαρμογή των τροπολογιών που προτείνετε αλλά η υποχρεωτική φύση είναι κάτι το οποίο στηρίζω. Ξέρω πως δεν συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι, γιατί στον πυλώνα 2 κάποια κρατημέλη κάνουν πολύ περισσότερα από άλλα. Όσον αφορά δε τη ρήτρα ενεργοποίηση του 2011, είμαι σίγουρος πως εννοείται πως θα μπορούσε να είναι 2009 ή 10 ή 11 και νομίζω πως το κείμενο πρέπει να ξεκαθαρίσει για την ευελιξία μεταξύ πυλώνων. Αναρωτιέμαι και πάλι τι άποψη θα είχαν οι αγρότες για το, να αποφασί... για το ότι αποφασίζουν τα κράτη-μέλη να πάρουν 20% από τον πυλώνα 1 και να το πάνε στον πυλώνα 2. Τι αντίκτυπο θα έχει στις πληρωμές τους και πώς θα χρησιμοποιήσουν την ευελιξία τα κράτη-μέλη. Είναι ανοιχτό το ζήτημα. Όσον αφορά τους ενεργούς αγρότες, δικαίως προσπαθείτε να αποφύγετε την πολυπλοκότητα της πρότασης της Κομισιόν για τη μέτρηση του εισοδήματος και τα λοιπά. Αν πάτε νομίζω σε μια σωστή κατεύθυνση. Η προσωπική μου άποψη εδώ πέρα είναι η εξή. Πρέπει να φροντίσουμε τα λεφτά να πάνε πράγματι σε ενεργούς αγρότες, αλλά είναι δύσκολο να έχουμε πανευρωπαϊκό ορισμό και τα κράτη-μέλη χρειάζονται κάποια ευελιξία αλλά και βεβαιότητα πως βεβαίως ε, δεν θα έχουν προβλήματα με τα μέτρα που θα λάβουν. Και υπάρχει ένας υφιστάμενος κανονισμός ο οποίος εάν το χρησιμοποιήσουμε σωστά μπορεί να εφαρμοστεί για να πηγαίνουν τα λεφτά στους ενεργούς αγρότες. Μετά κάποια σχόλια για τα μικρότερα αλλά εξίσου σημαντικά τμήματα του συστήματος για τις ε, μικρές εκμεταλλεύσεις πρέπει να είναι προαιρετικό, γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν καν να λάβουν μέρος. Κάποιες γενικές παρατηρήσεις για την απλοποίηση. Είχα υποσχεθεί πως δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, αλλά δεν νομίζω πως είναι απλό αυτό το μέτρο. Η αρχική πρόταση προσθέτει κόστος στα κράτη-μέλη, γραφειοκρατία και θα πρέπει να αποδείξουν ε, βεβαίω πώ θα κάνουν αυτά τα οποία του λέει η Κομισιόν και να ξοδέψουν χρήματα σε καιρούς δύσκολους. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε τα πράγματα πιο αποδεκτά και λιγότερο πολύπλοκα. Και βέβαια η μεγαλύτερη πολυπλοκότητα είναι να σταματήσουμε όλα τα δικαιώματα και να ξεκινήσουμε με ένα τελείως καινούριο σύστημα έχετε απομακρυνθεί από αυτή τη θέση, πρέπει να το ξαναδείτε, γιατί εκεί πέρα βρίσκεται η μεγαλύτερη δυσκολία για τα κράτη-μέλη. Οπότε, συνοψίζω λέγοντας πως υπάρχουν κάποια θετικά, πράγματι το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι κάπως πιο φιλοδόξο και όχι τόσο κοντά στην Κομισιόν. Είμαστε στην αρχή της διαδικασίας και πρέπει να ε, έχουμε ένα ευρύτερο όραμα ε, για την κοινή γεωργική πολιτική, λαμβάνοντα οπωσδήποτε πάντα υπόψη το τι σημαίνουν αυτά για τον κλάδο της γεωργίας και το να έχουμε μία βιώσιμη παραγωγή τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα προσφέρει ε, διατροφική ασφάλεια και βεβαίως ε, θα ανταποκρίνεται και στα ζητήματα του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ Μάριατ. Ο Τζορτζ Λάιον, μετά ο Τζιμ Νίκολσον Φυσικά, Τζιμ, μπορείς να μιλήσεις και για το δεύτερο πυλόν, αν θέλεις, γιατί εμείς ενώνουμε και τις δύο εκθέσεις. Ο Τζόρτ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω και εγώ την έκθεση του κυρίου Σάντος και τον ευχαριστώ για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε τις τελευταίες εβδομάδες και τον ευχαριστούμε που έλαβε υπόψη κάποιες από τις απόψεις που εκφράσαμε για τις άμεσες πληρωμές. Θα συμφωνήσω κάπως και με τις συνάδελφό λέγοντας πως η έκθεση την οποία δημοσιεύσατε δεν έχει κάποια φιλοδοξία, είμαστε πάρα πολύ κοντά προς την Κομισιόν. Πρέπει να είμαστε κάπως πιο φιλόδοξοι σε κάποιου για να έχουμε μια ισχυρή πολιτική θέση στι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Αλλιώ, τι θα καταλήξουμε, να είμαστε οπαδοί της Κομισιόν και να μην έχουμε δική μας θέση. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα όταν θα φτάσουμε στι τροπολογίε τώρα. Να αναφερθώ στα ζητήματα και να σχολιάσω σε αυτά. Πρώτα απ' όλα, το μεγαλύτερο και το δυσκολότερο είναι η αναδιανομή εντό των κρατών μελών. Και βεβαίω καλωσορίζω αυτό το οποίο είπατε για την εισαγωγή ενό μήνυμου με 65% κατά το οποίο κανένα κράτο μέλο δεν θα μπορεί να πέσει γιατί βεβαίως έτσι θα έχουμε ίδιε συνθήκε ανταγωνισμού υποψιάζομαι πως καθώς αυτό είναι ζήτημα βεβαίως διαπραγματεύσεων ε, του του δημοσιονομικού πλαισίου θα αποφασιστεί από τους αρχηγούς κρατών. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά οπωσδήποτε καλώς ορίζω την, προσπάθη, την κατεύθυνση προς την οποία πήγατε. Όσον αφορά την εσωτερική σύγκληση, εντό των κρατών μελών, είναι θετικό το ότι εξαιρέσατε τα κράτη-μέλη που ήδη χρησιμοποιούν το περιφερειακό αυτό μοντέλο δεν είναι ανάγκη να επανεφεύρουμε τον τροχό. Όσον αφορά την περίοδο αναφοράς ε, για την πιστοποίηση 2009-2011 θα πρέπει να ε, διευρύνουμε το δίχτυ για να μην ξεγλιστρήσει κανείς. Αλλά κάποιοι θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν ακόμα και με αυτά τα μέτρα. Θα δούμε τώρα αν χρειάζονται ειδικά μέτρα ή εάν το εθνικό απόθεμα θα το αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα αυτομάτως. Συμφωνώ με το ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα σε μια σύγκληση. Δεν ξέρω αν προχωράμε αρκετά, γιατί οπωσδήποτε η ισοπαίδωση αυτή του πρασινίσματος σημαίνει πως μιλάμε για ουσιαστική αναδιανομή στο πρώτο έτος όσον αφορά δε τη μείωση των προβλημάτων της αναδιανομής και το πώς θα το αντιμετωπίσουμε, συμφωνώ με τη γενική κατεύθυνση. Εγώ θεωρώ πως πρέπει να αυξήσουμε την περίοδο αυτή. Αν δούμε τα δύο παλαιά κρατημέλη που το κάνανε αυτό, τη σύγκληση, ε, χρειάστηκαν 7 χρόνια. Νομίζω πως αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς και να δούμε το εάν αυτό είναι το σωστό μοντέλο. Όταν μιλάμε για το πρασίνισμα, που είναι πάλι ένα από τα μεγάλα ζητήματα και εγώ θεωρώ πως χρειάζεται ένα μενού. Αυτό είχαμε ψηφίσει στην έκθεση DES. Αυτή ήταν η στάση της Επιτροπής μας, οπότε πρέπει να επιμείνουμε παρά την άρνηση της Κομισιόν να μετακινηθεί εδώ πέρα. Έχουν εντύπωση πως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να διαλέξουν από κάποια μέτρα. Αυτά δηλαδή τα οποία θα επηρεάσουν περισσότερο την περιοχή τους, την περιφερειά τους, γιατί σε πολλά κράτη-μέλη μέτρα βιοπικιλότητας υπάρχουν ήδη και εφαρμόζονται. Χρειαζόμαστε ζητήματα, μέτρα που αντιμετωπίζουν την ε, κλιματική αλλαγή και την καλύτερη χρήση των ε, διαφόρων πόρων. Οπότε θα πρέπει νομίζω να φροντίσουμε να γίνει κάτι τέτοιο στη φάση των τροπολογιών. Καλώ ορίζω επίσης το ότι κάποιε από τις αλλαγέ των τριών μέτρων του πρασινίσματος που είναι κάτι το οποίο θα εξετάσουμε και θα δούμε εάν μπορούν να λειτουργήσουν πρακτικά. Επίσης καλωσορίζω την πιθανότητα του να μπουν σε κάποια πιστοποιημένα συστήματα αγρότες και μετά αυτομάτως να θεωρείται πως συμμορφώνονται με τις απαιτήσει πρασινίσματος. Η ανησυχία μου είναι πως περιορίζεται στα ίδια μέτρα που είναι πάλι τύπου βιοπικιλότητας και νομίζω πως αυτό είναι το μεγάλο μειονέκτημα, ότι έχουμε κολλήσει στη βιοπικιλότητα αποκλείοντας τα μέτρα της κλιματικής αλλαγής. που κατά την άποψή μου είναι λανθασμένη άποψη. Πρέπει να δώσουμε στα κράτη-μέλη και τις περιφερειές την ευκαιρία να διαλέξουν εάν είναι μέτρα βιοπικιλότητας ή αυτά που αφορούν την κλιματική αλλαγή. Οπότε θα ήθελα έναν ευρύτερο ορισμό. Πανεργός αγρότης ε, πράγματι νομίζω όλοι αντιλαμβάνονται πω δεν τίθεται ζήτημα εισοδήματο κτλ. Θα δούμε τώρα το τι θα επιτραπεί στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν. Εγώ θα ήθελα, δεν ξέρω το πώς θεωρείτε ότι μπορεί να δουλέψει αυτό που λέτε με το μη ενεργό γεωκτήμονα κτλ. Όσον αφορά δε, το, το πλαφόν θα δούμε κάποιες εναλλακτικέ λύσεις και πάλι ανισχώ εδώ πέρα για την ευελιξία μεταξύ πυλώνων, ε, την ε, δυνατότητα μεταφοράς του 20%. Ξέρω πως είναι πορτογαλικό ζήτημα και στο Ηνωμένο Βασίλειο υφίσταται Ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη ρύθμιση για τα ζητήματα της ε, ανάπτυξης υπαίθρου. Συνολικά η έκθεσή σας μας πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω πως αυτό το οποίο πρέπει να κάνει το Κοινοβούλιο να είναι πολύ πιο φιλόδοξο για να έχουμε μια σαφή πολιτική θέση όταν θα πάμε στις διαπραγματεύσεις. Πρέπει να θυμόμαστε πως δεν προσπαθούμε εδώ πέρα να τα γράψουμε όλα οριστικά. Θέλουμε μια ισχυρή πολιτική θέση, μια αρχική διαπραγματευτική θέση για να μπορούμε να κάνουμε και κάποιες ε, διαπραγματεύσεις. Εγώ φοβάμαι πως είμαστε πάρα πολύ κοντά στην Κομισιόν. Και καταλήγουμε υποστηρικτές ε, κάποιο άλλο αντί για παίκτες. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ Τζόρτζο. Συνεχίζουμε. Ο Τζιμ Νίκολσον και μετά Μάρτιν Χάουσλινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για όλες τις προτάσεις που κάνει. Όπως ε, είπε και ο ίδιος, είναι αλληλένδετες και αλληλοσυμπληρούμενες. Ε, και όσο περνάει ο καιρός, οι μέρες, οι μήνες, θα διαπιστώσουμε ποια διάσταση απόψεων υπάρχει και αν υπάρχει μέσα στο Κοινοβούλιο. Για την έννοια του ε, ενεργού γεωργού δεν πρέπει να ακολουθήσουμε τον δρόμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρέπει να ακολουθήσουμε τον αρνητικό κατάλογο και όπως είπαν και κάποιοι θα, ίσως υπάρχουν ήδη διαθέσιμες πολιτικές που μπορούμε να εφαρμόσουμε ούτως ώστε να είναι εύκολο να στοιχειοθετηθεί ποιος είναι ενεργός γεωργός και να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί που δουλεύουν την Αγή και παράγουν, αυτοί θα θεωρούνται ενεργοί γεωργοί. Θέλω να πω ότι αντιτίθεμαι ε, κάθετα ε, προς τις στις θέσεις του εισηγητή ως προς ε, το προσδιορισμό του ανώτατου ορίου. Θα πολεμήσω μέχρι τελικής επτώσης κατά του ανώτατου ορίου. Πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνουν όσο έχουν οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, διότι ε, όντω ε, θα πρέπει να ξέρουμε πόσοι δουλεύουν τη γη, πόσοι είναι μέσα στην γεωργική εκμετάλλευση, τι μέγεθο έχει, αλλά κυρίω όχι αυτά που μα προτείνει εδώ η συγγετής. Ε, για αυτέ τι προτάσει. Τι πιστεύω. Πιστεύω ότι παρά είναι, ε, προσεγγίζουν υπερβολικά τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, δεν θέλουμε ημίμετρα, δεν θέλουμε μια ημιτελή θέση. Ε, χρειαζόμαστε μια ξεκάθαρη θέση και ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη θέση τη δική μας και τη θέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί έτσι θα έχουμε ουσιαστικέ διαπραγματεύσεις, όχι να πηγαίνουμε λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά, λέμε τα ίδια. αντί να πρασινίσουμε το δεύτερο πυλώνα, ε, πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό, αλλιώς θα έχουμε υπερβολική και ακόμη περισσότερη ε, γραφειοκρατία χτες. Ε, είδαμε ότι μπορεί να προκύψει μείωση της ε, γραφειοκρατίας με την έκθεση Λαβία. Εδώ το αντίθετο συμβαίνει. Θα ε, στραγγαλίσουμε περισσότερο τη Γεωργία και τους Γεωργούς ε, με τόση πολλή γραφειοκρατία, με όλα αυτά που τους ζητούμε σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Αυτή η εστίαση στο μικρό Γεωργό. Εντάξει, αλλά γιατί όμως όχι και για το μεγάλο το Γεωργό. Αφού έχουμε και από τους δύο, έχουμε και μικρούς, έχουμε και μεγάλους και όλους πρέπει να τους βοηθήσουμε. Δεν μπορούμε να ξεχωρίζουμε έτσι τους Γιώργους. Πρέπει να επιβιώσουν όλοι, γιατί όλοι τροφή παράγουν. Και όλοι εργάζονται ιδιαίτερα σκληρά. Λοιπόν, για το θέμα του μενού. Ξέρω, δεν αρέσει αυτή η λέξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ όμως καμία αμφιβολία δεν έχω. Στο τέλος ε, θα παραμείνει το μενού. Ε, δεν ξέρουμε απλώ σε ποια μορφή. Α αρχίσουμε λοιπόν ήδη τη συζήτηση για το πώ θα διαμορφωθεί. Τι έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μα λέει ότι αποκλείεται. Εγώ του λέω τώρα ότι θα συμβεί. Αυτό πρέπει να συμβεί. Αυτό χρειαζόμαστε. Αν θέλουμε να λειτουργήσουν αισίω ε, πολλέ από τι νέε προτάσει. Και πρέπει να πω και κάτι άλλο εδώ. Μιλάμε για την ενιαία ενίσχυση και τι συμβαίνει στα διάφορα κράτη-μέλη ε, και μιλάμε για την περίοδο από το 1998 στο 2002 με τη, τα ιστορι, τις ιστορικές αναφορές. Δηλαδή μιλάμε ε, για ε, εκμεταλλεύσεις εκτροφής ε, διαφόρων ζώων και οι ενισχύσει που πήγαιναν σε αυτές τις εκμεταλλεύσεις μεταφέρονται τώρα σε εκμεταλλεύσεις, σε λεόνες, σε γαλακτοκομικές μονάδες λέγοντας ότι προστατεύουμε τη γεωργία, αλλά τελικά δεν προστατεύουμε τα εγωπρόβατα. Προσοχή! διότι ε, θα ε, περιέλθουν αυτοί οι δύο τομείς ε, της γεωργίας σε ακόμη δυσχερέστερη θέση και στην περιοχή μου μειώνονται οι πληθυσμοί στα εγωπρόβατα και δεν βλέπω πώς θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Το ο εισηγητής ε, προσπαθεί να λύσει επίση το πρόβλημα του νέου γεωργού ε, και μας λέει ότι ίσω πρέπει να χρηματοδοτούμε και την ε, μίσθωση της γης, τη χρονομίσθωση. Ίσως και να λειτουργήσει αυτό το σύστημα, αλλά αν χρηματοδοτείται κατά αυτόν τον τρόπο την γεωργική εκμετάλλευση θα ανέβει η τιμή ε, του αγροτεμαχίου και θα ε, ε παλεύουν όλοι μεταξύ τους ε, και θα επικρατήσει αυτός που έχει τα περισσότερα λεφτά για να πληρώσει το τίμημα. Ο νέος γεωργός θα πρέπει ε, όταν είναι έτοιμος να κάνει την αλλαγή στη ζωή του και να ασχοληθεί με αυτή την γεωργική δραστηριότητα ε, να μπορέσει να έχει τα απαιτούμενα μέσα και σωστά αυτά που λέτε για ε, τους παλιούς γεωργούς, αλλά σε καμία περίπτωση το νέο σύστημα δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικό, γιατί τα νέα κρατημέλη αποκλείεται ε, να ακολουθήσουν αυτό και να εφαρμόσουν αυτό το νέο καθεστώς, ε, κυρίως γιατί δεν θα έχουν την απαιτούμενη χρηματοδότηση. Βρίσκω πολύ ενσυχητική αυτή την πρόταση. Επίσης, μιλάτε για τα κράτη-μέλη που για το δεύτερο πυλώνα για το πρασίνισμα θα εφαρμόσουν αυτό το ποσοστό του 30%. Πολύ πολύ ωραία αυτά, αλλά τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε τα χείριστα δυνατά κονδύλια διαθέσιμα για το πυλώνα 2 και μόνο με την πολλαπλή μορφος, ή μάλλον με την... Ε, με την προσαρμογή, την αναπροσαρμογή των ποσών θα καταφέρουμε να βοηθήσουμε την γεωργία γιατί ε, είναι ήδη πάρα πολύ χαμηλά τα ποσοστά του εθνικού μας αποθέματος που προβλέπονται για το δεύτερο κονδύλιο. Θα, δεν ξέρω ακριβώς με ποιο τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε πιο αποτελεσματικά την κατάσταση. Πολλοί έχουν έτοιμες λύσεις, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι προσχήματα και δεν πρέπει να θεωρούμε ότι οι άνθρωποι επιτόπου θα μπορέσουν εύκολα να εφαρμόσουν όλα αυτά τα νέα συστήματα. Ε, δεν συμφωνώ με όλα αυτά τα στοιχεία που προτείνει ο εισηγητής, γιατί θεωρώ ότι αν εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα δεν θα λειτουργήσουν στην πράξη. Ε, κατά τη διάρκεια λοιπόν της εξέτασης του ζητήματος από την Επιτροπή μας ε, θα πρέπει να μην παραγνωρίζουμε τη σημασία των ε, βασικότερων μεγεθών και της πραγματικότητας που ισχύει στα διάφορα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστούμε Τζιμ, τώρα Μάρτιν Όσλιν και στη συνέχεια Άγνιο παρακαλώ. Ναι. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις, δεν ελήφθησαν όλες υπόψη, ελπίζουμε παραπέρα στις διαπραγματεύσεις να συμπεριληφθούν. Έγινε πολλή λόγος για το ότι το θέμα είναι να είμαστε φιλόδοξοι, πιο φιλόδοξοι από την Κομισιόν. Η φιλοδοξία πάει σε λάθος κατεύθυνση όμως. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε αυτό το οποίο λέει η Κομισιόν, μια νέα αιτιολόγηση για τις πληρωμές, δηλαδή κλιματική αλλαγή για να δώσει τα λεφτά ο φορολογούμενος. Δυστυχώς εδώ σε πάρα πολλά σημεία πάμε στη, στη, σε άλλη κατεύθυνση. Να επεκταθεί το σύστημα, δηλαδή να συνεχίσουμε να πληρώνουμε για μία υφόρο γεωργία. Εκεί πέρα είναι η κριτική μας. Αν δείτε τις προτάσεις, ναι, εντάξει, υπάρχει απλοποίηση, σε κάποια συμφωνούμε, αλλά αν έχουμε απλοποίηση εις βάρος των περιβαλλοντικών μέτρων, τότε είμαστε πολύ επικριτικοί. Στο σημείο δε της ε, αλλαγής ε, καλλιεργειών ε, και Κομισιόν περιορίζεται σε ένα 70% και δεν μας βοηθάει πάρα πολύ. Εμείς θέλουμε μια πραγματική αλλαγή καλλιεργειών και αμύψη σπορά και έλεγχο. Όταν λένε πως δεν ελέγχονται αυτά τα πράγματα, δεν είναι δυνατόν. Μια χαρά ελέγχονται. Και οπωσδήποτε αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο αποδίδει. Πρέπει να κάνουμε κάτι κατά της ε, Μονοκαλλιέργεια ε, αυτό το οποίο βλέπουμε με τις εκτάσεις καλαμποκιού. Όσον αφορά δε τις εκτάσει. εκτάσεις, ε, χαιρετίζουμε όλη την πρόταση της ε, Κομισιόν, αλλά η ημερομηνία έναρξης μεταρρύθμισης νομίζω είναι λαθασμένη και οπωσδήποτε θα πρέπει να λάβουμε τώρα μέτρα. για τις συγκεκριμένες προτάσεις τώρα του πρασινίσματος. Εάν προτείνει ο εισηγητής ε, κάποια απλοποίηση, ναι εντάξει και στις μικρότερες εκμεταλλεύσεις συζητάμε και στη Γερμανία ε, το να τις εξαιρέσουμε, αλλά αυτό, μιλάει, αυτό σημαίνει στη Γερμανία 50% των εκμεταλλεύσεων και 80% στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι πολλές ήδη. Αν, αν το πάμε δε και με το στρεματικό κριτήριο, τότε 20% των εκτάσεων δεν θα έχουν καθόλου τέτοια μέτρα πρασινίσματος. Τότε τι σημαίνει αυτό, εάν δεν έχουν το 7% οι μικρότερες εκμεταλλεύσεις, οι μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις πρέπει να κάνουν περισσότερα. Δηλαδή, αλλιώς θα μπορούσαμε να το μοιράσουμε με ένα όριο τα 100 εκτάρια, αλλά να το αλλάξουμε τόσο πολύ ώστε να μην απομείνει στο τέλος ε, παραελάχιστο, το ζήτημα είναι τι, τι, τι απομένει από αυτό το πρασίνισμα. Καμία μη ψησπορά, καθόλου περιοχές ε, οικολογικής προτεραιότητας, οπότε θα αναρωτηθεί και το κοινό ποια είναι η νέα κατεύθυνση. Πού είναι η αηφορία, εκεί πάμε ή πάμε για προστασία του status quo. Εάν λοιπόν υποθέσουμε πως ε, ε, και οι μόνιμες καλλιέργειες θα, θα λάβουν μέτρα, βεβαίως αυτό είναι κάτι το λογικό και υπάρχει κάτι το οποίο, στο οποίο ασκήσαμε και χτες κριτική αυτό το 13%, το 30% με του προσθενίσματος. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε τελείως εθελοντικό. Πρέπει να το συνδέσουμε με το 70% των πληρωμών. Δεν θα γίνει τίποτα. Θα μας πούνε πως... Ε, ε ξέρετε τι θα γίνει. Θα πάρουν το 70% των πληρωμών, θα συνεχίσουν την εντατική γεωργία και δεν θα γίνει τίποτα. Πρέπει να υπάρξει μια σύνδεση μεταξύ του 30% πρασινίσματος και 70% βασικής πληρωμής, αλλιώς δεν θα λειτουργήσει τίποτα. Και δεν μπορούμε να δίνουμε λεφτά για μία εφόρο γεωργία. Αυτή είναι μεγάλη, νομίζω, διαφορά μεταξύ των όσων προτείνει ο ε, εισηγητής και των όσων προτείνουμε εμείς. Επίσης ο κύριος Νίκολσον που λέει θα υπάρξει μενού. Όχι, εμείς ε, δεν το θέλουμε αυτό. Το να έχουμε μενού τώρα για το πρασίνισμα ε, Εκεί πέρα είναι ένα κουτί από το οποίο δεν ξέρουμε τι θα ξεπηδήσει μέσα. Και δίνουμε το ελεύθερο στα κράτη-μέλη να κάνουν ό,τι θέλουν. Εκεί πέρα έχω τις αμφιβολίες μου αν θα το κάνουν τόσο σοβαρά. Αν δούμε και την αντίστασή τους κατά του πρασινίσματος. Οπότε θα προτιμούσα να μην έχουμε μενού ε, όπου θα διαλέγει ο καθένας ό,τι θέλει. Γιατί πρέπει να υπάρχει μια αξιοπιστία τελικά αυτής της μεταρρύθμισης. Θεωρώ στους ορισμούς τι είναι ο, τώρα, ο ενεργός γεωργός Έχουμε πει πως πρέπει να γίνει ο κατάλογος αρνητικός να πούμε τι δεν είναι δηλαδή ένα ενεργός αγρότης, αλλά βέβαια δεν είναι ακόμα οριστικός αυτός εδώ ο κατάλογος, πρέπει να συμπληρωθεί. Πρέπει λοιπόν να επεκταθεί και θα κάνουμε τις ανάλογες προτάσεις τώρα. Κατά την άποψή μα και εδώ πέρα είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για μα. γιατί είναι κάτι το οποίο πάει τελείως ε, στην κατεύθυνση. Να πληρώνουμε 435.000 ευρώ μια εκμετάλλευση η οποία βγαίνει εκτός παραγωγής. Γιατί δηλαδή θέλουμε να βοηθήσουμε τις μικρές επιχειρήσεις, το μικρό αγρότη και μετά 35.000 ευρώ για να βγει και μετά 35.000 ευρώ για να βγει κάποιος εκτός παραγωγής, όχι είναι τελείως αντιπαραγωγικό και μετά λέτε ότι προωθούμε έτσι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Μα τι κάνουμε, ε, βοηθάμε το μικρό αγρότη ή θέμε να τον εξαγοράσουμε για να φύγει εκτός παραγωγής, τι από τα δύο κάνουμε. Σε πολλές ε, περιοχές ε, για τη Γεωργία για τους γεωργούς δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα βιοπορισμού. Οπότε να τους λέμε βγες εκτός παραγωγής είναι λανθασμένο. Για το πλαφόν ο συγκητής πρότεινε να γίνει πιο έντονο αυτό. Αλλά από αλλού θέλει να το χαλαρώσει. Συνεταιρισμοί τώρα να εξαιρεθούν από το πλαφόν. Εντάξει, είναι μια σκέψη, αλλά όλοι ξαφνικά θα βρεθούν ε, Εντό συνεταιρισμών και δεν θα αφορά κανέναν μετά το πλαφόν. Και η Κομισιόν εδώ πέρα το βλέπει με κάποια ε, συμπάθεια. Νομίζω πως ε, όμως η πρόταση της Κομισιόν είναι πιο λογική από το να λέμε πως εκ των προτέρων εξαιρούνται όλοι οι συνεταιρισμοί. Δηλαδή στην Ανατολική Γερμανία ε, δεν θα αφορά κανέναν αυτό το μέτρο, έτσι, γιατί είναι όλοι σε συνεταιρισμό. Η Verteilung zwischen den Mitgliedstaaten ist, glaube ich, äh, ein richtiger Ansatz gewählt worden. Da sind wir auch dabei. Wir müssen. Οπότε. Βεβαίω, ω ζήτημα του περιβάλλοντο πρέπει να δούμε και το θέμα τη δικαιοσύνη εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αν υπάρχει αυτή η προσέγγιση δεν μπορώ να το κρίνω. Και πρέπει να δούμε μαζί πρώτο και δεύτερο πυλώνα και βεβαίως ε, η μεταφορά αυτή από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα έχει κάποιο νόημα, δίνει ευελιξία στα κράτη-μέλη, αλλά όχι αντιστρόφως, όχι από το δεύτερο στον πρώτο. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε, είναι σαφές. Και πρέπει να δώσουμε βεβαίως και στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα χρηματοδότησης ε, από πρώτο στο δεύτερο πυλώνα, αλλά όχι αντιστροφή. Λοιπόν, αυτά ω μια πρώτη τοποθέτηση. Πρέπει να έχω ξεχάσει και κάποια πράγματα, αλλά έχουμε ούτω ή άλλω καιρό μπροστά μα. Ε, κάτι άλλο να πω θετικό, πω ο εισηγητή συμπεριέλαβε και τα πρωτεϊνούχα φυτά. Θα υπάρχει πρόταση στη Γερμανία να πούμε ένα 15% ε, με ένα μίνιμουμ, αλλά εν πάση περιπτώσει χαιρετίζουμε το ότι έχουμε τα πρωτεϊνούχα φυτά και συμπεριλαμβάνονται. Οπότε υπάρχουν θετικές ε, προσεγγίσεις και αρνητικές. Πρέπει λοιπόν να βρούμε εδώ πέρα μια διέξο. Οπότε έχουμε την ε, δυνατότητα και πρέπει να έχουμε τη φιλοδοξία να πάμε σε μια πορεία πιο φιλοδοξία από την οποία θέλει η Κομισιόν και να μην τα αφήνουμε τελείως στην επιλογή των κρατών. Να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα συνεπέ πρασίνισμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ Μάρτιν. Ο Άγνιου και μετά ο Βασιβόφσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι αδύνατο το καθήκον που αναθέσαμε στον εισηγητή. Για να δούμε κάποια, κάποιες από τις επικεφαλίδες. Ενεργός γεωργός. Μα το κράτος μέλος πρέπει να αποφασίσει σίγουρα πράγματα και πρέπει να βασίζεται η απόφαση στο αν ε, υπάρχει κίνδυνος ε, ως προς ε, την οικονομία για την εκμετάλλευση. Δηλαδή όταν λαμβάνει κάποιος μια ενίσχυση και θεωρεί ότι το κράτος μέλος είναι οριακή κατάσταση για κάποιον, λοιπόν να του ζητήσει να αποδείξουν τι παράγει η εκμετάλλευση. Είναι ενεργή η γεωργή. αντί να επενδύουμε και να χάνουμε τα λεφτά μας διότι η έκταση είναι επιλέξιμη. Απλά είναι τα πράγματα επίσης. Ε, ε, θεωρώ ότι με το που θα αποφασίσει η χώρα μου δεν μπορεί να πηγαίνει ο γεωργός ε, υπονομεύοντας την εθνική απόφαση ε, να προσφύγει στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ε, γης που δεν είναι επιλέξιμος μας λέει ο εισηγητής. Και πάλι η απόφαση του κράτους μέλους πρέπει να είναι αυτό και οποιοδήποτε πλεόνασμα έχουμε αν δηλαδή δεν επιδοτηθεί μία περιοχή λοιπόν θα πρέπει να μπαίνει στο εθνικό απόθεμα για τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών μάλιστα. Ε, ακολουθείτε Ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση ο εισηγητή, αλλά πραγματικά κυρίω για τη χώρα μόνο αναρωτιέμαι γιατί το χρειαζόμαστε αυτό. Οι ε, μονοκαλλιέργειε σπάνια ε, απαντώνται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτοί και αυτοί που επιλέγουν τη μονοκαλλιέργεια ακολουθούν και περιβαλλοντικά φιλικά ε, καθεστώτα, δηλαδή ε, ε, φιλικές προς το περιβάλλον γεωπονικές μεθόδους. Οπότε δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει για τις περιοχές οικολογικής εστίασης θεωρώ ότι αυτό το μέτρο θα μπορεί να θεωρηθεί και ως αγρανάπαυση ουσιαστικά. Και γιατί λοιπόν να μην επιτύχουμε με ένα σπάρο δύο τριγώνια, διότι Μα λέτε εσεί ότι πρέπει όταν έχει κάποιο δύο καλλιέργειε ε, πρέπει να βρει και μία τρίτη ε, για να πιάσει το 75%. Ο μελισσοκόμο όμω. Ε, δεν έχει το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή ορισμένοι μπορούν να θεωρήσουν αυτό το σύστημα επιδότησης είναι η κρυφή επιδότηση για, τους, για τα πρωτεϊνούχα φύτα. λοιπόν, Ξέρετε ότι για κάθε... Ε, δεν έχουμε μεγάλη απόδοση ως προς τα χρήματα που δίνει η χώρα μου ε, στην ε, κυνηγιορική πολιτική, οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί είναι στο προσυμφέρον της χώρας μας να το κάνουμε αυτό. Σε σχέση τώρα με τον νεαρό γεωργό, νομίζω ότι απλώς θα συνεχίσουν τα παιδιά των γεωργών να καλλιεργούν τη γη. Δεν πιστεύω ότι θα έρθει νέο αίμα και με τις νέες ρυθμίσεις δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια σημαντική διαφορά και πρέπει να είναι προαιρετικό το σύστημα. Διαφωνώ με κάποιους συναδέλφους για να έχετε νέο αίμα χρειάζεστε υποτροφίες. Ε, ε, πέρα από τον αρνητικό κατάλογο ε, πρέπει να επιλεγούν από το κράτος κάποιοι άνθρωποι για λόγους κοινωνικής κινητικότητας που θα υποστηριχθούν από το κράτος για να αρχίσουν να ασκούν τη γεωργική δραστηριότητα. Ούτως ή άλλως για τους μικροκαλλιεργητές πρέπει να είναι ε, προαιρετικό το σύστημα. Ε, ε, φυσικά τώρα με 28 χώρες είναι εξαιρετικά περίπλοκα όλα αυτά τα ζητήματα και εγώ δεν θέλω να χάνουμε τα χρήματα των φορολογουμένων με τη φενάκι που μας προτείνει ότι δηλαδή θα δεσμεύουμε και το άζωτο με τις νέες καλλιέργειες ε, εγώ πιστεύω ότι οι παραδοσιακοί ε, γεωργοί και <coughs> εκτροφείς θα σοκαριστούν με το νέο σύστημα που ε, προτείνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρος πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τον εισηγητή τον κύριο Κάπουλα Σάντος ε, για τη δουλειά του και για την προσπάθεια στην προετοιμασία της έκθεσης που φυσικά τίνει προς την σωστή κατεύθυνση. Εγώ τον υποστηρίζω 100% αλλά θα ήθελα να αναφέρω κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο και αποτελεί και το πιο δύσκολο σημείο, δηλαδή τη διανομή των πληρωμών. Πρέπει να θυμίσουμε ότι εμείς δεν κάνουμε μόνο πολιτική, αλλά και είμαστε και νομοθέτες πέρα από πολιτική. Έχουμε εδώ ένα νομοθετικό ψήφισμα, το οποίο θα γίνει νόμος, οπότε πρέπει να θυμίσουμε τους βασικούς κανόνες που ισχύουν εδώ και που λένε σαφώς ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία διάκριση κανενός σε όλη την Ένωση λόγω υπηκότητας, δεν πρέπει να υπάρχει δηλαδή, να υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ παραγωγών και προϊόντων στα κράτη-μέλη. Πρέπει εμείς στην εφαρμογή της ΚΑΠ να λάβουμε υπόψη τις περιφερειακές διαφορές, αλλά όχι τις διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Δεν μπορούμε εμείς να διαφοροποιούμαστε έναντι πολιτών συγκεκριμένων χωρών στη βάση της ηθαγένειας. οι διαφορές μειώνονται εν μέρη, διότι η πρόταση της Κομισιόν είναι αυτή, αλλά υπάρχουν τεράστιες διαφορές και δυσκολίες. Έχουμε δύο χώρες, μια παλιά χώρα, η Δανία, και μια νέα χώρα, η Λιθουανία, που γεωγραφικά ανήκουν στην ίδια περιφέρεια και έχουν 2.600 εκτάρια πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. 900 εκατομμύρια θα πάρει η Δανία, ενώ η Λιθουανία μόνο 450. Το μισό. Και αυτό στα τέλη της περίοδου, γιατί σήμερα η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη. μισό δις ευρώ λοιπόν μισό συγγνώμη εκατομμύριο ευρώ πάει μόνο σε μία χώρα και θα καταστρέψει την Λιθουανική Γεωργία όπου σίγουρα το κόστος είναι διαφορετικό αλλά οι γεωργοί δεν διαφέρουν δεν διαφέρει η τιμή των ε, τρακτέρ και των αγροτικών μηχανημάτων ε, ούτε των φυτοφαρμάκων. Οι γεωργοί πάνε στη Γερμανία για να αγοράσουν και τα μηχανήματα και τα λοιπάσματα. Δηλαδή και αν το δούμε ιστορικά τι σημαίνει. Σημαίνει ότι κάποιοι θα πάρουν λεφτά, γιατί πάντα παίρνουν λεφτά, ιστορικά, και άλλοι λιγότερα γιατί πάντα ιστορικά παίρναν λιγότερα. Λοιπόν αυτού του είδους η φιλοσοφία δεν πρέπει να συνεχίσει να ισχύει, πρέπει να σταματήσει διότι δεν σέβεται τις συνθήκες και πρέπει να καταργηθεί. Θέλω να θυμίσω στους παρόντες ότι Δεν μπορούμε από τους εθνικούς προϋπολογισμούς να παίρνουμε χρήματα για να χρηματοδοτούμε μόνο μία ευρωπαϊκή χώρα από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Καταλαβαίνω ότι μία μείωση των πληρωμών για ορισμένες χώρες θα ήταν απαράδεκτη. Αλλά ας συνεχίσουν να πληρώνουν παίρνοντας ένα μεγαλύτερο κομμάτι χρηματοδότησης από το δικό τους προϋπολογισμό. Αν κάτι είναι λιγότερο άδικο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι άδικο. Και το πρόβλημα, το οποίο το λύσαμε εμείς στη χώρα μας, φαίνεται να εντείνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας εστίες κρίσης που θα ενισχυθούν από τη διαφορά αυτών των πληρωμών. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από την απόδοση μερικής δικαιοσύνης. Η Ελίζα Κόστιγκερ και μετά ο Πόλσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή μας τον Λούις Κάπουλας για τη δουλειά που έχει κάνει και για την δυνατότητα που έδωσε στους ε, σκιώδεις να συμμετάσχουν διαβάζοντας ε, τις τροπολογίες του εισηγητή αμέσως προέκυψε μία ερώτηση ο εισηγητής εδώ πέρα χρησιμοποιεί συχνά τον όρο ε, λυπή γεωργοί, λοιποί εργαζόμενοι και εκμεταλλευτές ε, γης. Ποιοι είναι αυτοί οι λοιποί γεωργοί, δεν καταλαβαίνω, ποιοι θα μπορούσαν να στηριχθούν από τα προγράμματα ανάπτυξης υπαίθρου. Επίσης, ε, όταν μιλάμε για τις άμεσες πληρωμές του πρώτου πυλώνα, θα πρέπει να ορίσουμε το τι σημαίνει ενεργός γεωργός μέσω μια οπωσδήποτε δημόσια συζήτηση, η οποία μας έχει πει πως θα πρέπει να ενισχύσουμε ακριβώς όσου πραγματικά συμμετέχουν στην παραγωγή. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα σαφής ορισμός για να μην ε, προσπαθούμε μετά να δικαιολογούμε τα δικαιολόγητα. Οπότε χαιρετίζω την πρόταση του εισηγητή όσον αφορά τα γεωργο περιβαλλοντικά εκεί πέρα που λέει πως τουλάχιστον 13% ε, θα πρέπει να πάνε για ε, τέτοια μέτρα ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτό το οποίο είχαμε θέσει ως στόχο της ε, μεταρρύθμισης δηλαδή να υπάρξει μια οικολογική μεταρρύθμιση η κυρία Μαγκίνες ήδη αναφέρθηκε σε μια βασική πληρωμή, δηλαδή τη συζήτηση που προκύπτει από όλο αυτό το ζήτημα, για τις βιολογικές καλλιέργειες νομίζω και εκμεταλλεύσεις υπάρχει μια διατύπωση στο οποία δεν διαφωνεί κανένας. Οπότε θα ήθελα εδώ πέρα να υπενθυμίσω πως ε, οι πιστοποιημένες ε, εκμεταλλεύσεις με τα σχετικά προγράμματα που υπάρχουν σε πολλά κατημέλη δεν θα πρέπει να βρεθούν ξαφνικά αδικημένες, ιδίως ε, όταν μιλάμε για βιολογική γεωργία, γιατί ναι. ήδη σε πάρα πολλές χώρες έχουν γίνει πάρα πολλά, τα οποία ήδη βρίσκονται και πάνε παραπέρα από το δικό μας το πρασίνισμα. Κάτι άλλο επίσης ο συναδελφός έννοιο αναφέρθηκε. Ο κύριος Άγνιο με συγχωρείτε, βεβαίως αναφέρθηκε στο πρασίνισμα κτλ να πω πως ε, πολύ απλά ε, για το νέο αίμα και τη νέα γενιά δεν ανάγκη να πάει στο γιο, υπάρχουν και κόρες. Και πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι γυναίκες εδώ πέρα, γιατί θεωρώ πως οι γυναίκες στη Γεωργία κάνουν πάρα πολλά. Και οπωσδήποτε θα πρέπει να συνεχίσουμε να το αναφέρουμε αυτό, να διαθέτουμε πράγματι τα ορθά μετά στη διάθεσή του. Όσον αφορά τώρα την ε, αναδιάρθρωση αυτή και τις πληρωμές ε, για πέντε έτη για την αναδιάρθρωση, εγώ θέλω να αναφερθώ στο πρόβλημα ε, που θα υπάρξει αν έχουμε προβλήματα στον υπολογισμό και στους ελέγχους ε, πως ε, πάρα πολύ συχνά υπάρχει ο κίνδυνος ε, για τους γεωργούς, πως τα πέντε χρόνια σημαίνει πως στο τέλος μπορεί να χρειαστεί να επιστρέψουν ένα πάρα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, οπότε θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ενέχουμε εις βάθος. Όσον αφορά την ε, δυνατότητα στήριξης επενδύσεων ε, ε, που θα λαμβάνουν υπόψη και την προστασία των ζώων και την φωτοπροστασία είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι θα πρέπει να έχουμε ίδιες συνθήκες εντός της Ευρώπης και αν είναι να γίνονται αλλαγές τότε οι γεωργοί σε όλη την Ευρώπη πρέπει να έχουν την ίδια στήριξη παντού για τη συμπερίληψη της ε, δασοκομείας ε, χαιρετίζω την πρόταση του εισηγητή αλλά θα πρέπει να δούμε τότε και το ζήτημα της ε, εφορίας, ειδικά όσον αφορά τους στόχους του 2020. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στον τομέα της και στην ενέργεια και στην προστασία του κλίματος. Νομίζω πως μπορούμε εδώ πέρα να τα συμπεριλάβουμε αυτά. Οι μειονεκτικές περιοχές αναφέρθηκαν ήδη. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το ότι εδώ πέρα συμπεριέλαβε τις προτάσεις μας για τη διαγραφή του άρθρου της Κομισιόν. Εγώ θα ήθελα να αναφερθούμε πολύ περισσότερο στην έκθεση Dorfman που ούτως ή άλλως έχει εγκριθεί Γι' αυτό θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό η ημερομηνία αυτή που πρότεινε ο εισηγητής να γίνει δεκτή και θεωρώ πως οπωσδήποτε το κοινοβούλιο θα πρέπει να τα διαθάλα. αλλά βεβαίως δεν γίνεται αυτό με τη σημερινή με τι σημερινέ επιστημονικέ γνώσει όσον αφορά τη διαχείριση του κινδύνου βλέπω κάπω επιφυλακτικά τι προτάσει της ε, Κομισιόν και του εισηγητή για χώρες οι οποίες τώρα δεν τα καταφέρνουν είναι πάρα πολύ δύσκολο να χρηματοδοτήσουν αυτά τα μέτρα όπως προτείνονται αυτή τη στιγμή από την Κομισιόν ε, ή για χώρες οι οποίες ε, χρησιμοποίησαν το άρθρο 68 για τις άμεσες πληρωμές που τους έδινε κάποιες δυνατότητες. Θεωρώ λοιπόν πως πρέπει να γίνει, είναι θετικό το ότι προτείνει μια αξιολόγηση αυτών των μέτρων ο εισηγητής, αλλά επίσης θα πρέπει ως ε, Επιτροπή Γεωργίας να ρίξουμε μια ματιά στο πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτόν τον τομέα. Για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης υπαίθρου και το προτινόμενο παράδειγμα του εισηγητή. Χαιρετίζω την προσέγγιση η οποία επιλέχθηκε για την κατανομή. Να πάμε δηλαδή σε ένα μέσο όρο κάποιων περίοδων, όχι μόνο ένα συγκεκριμένο έτος. Είναι σημαντικό, θεωρώ πως η Κομισιόν έχει κάνει λάθος. Αν πάρουμε μόνο το 2013 ως έτος αναφοράς, δεν είναι νομίζω μια σωστή εικόνα των όσων γίνονται σε σειρά ετών στη χρηματοδότηση της κοινή γεωργικής πολιτική. Κάτι άλλο το οποίο δεν ανέφερε ο εισηγητή, αλλά εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό είναι οι προτινόμενε αλλαγέ στο ποσοστό συγχρηματοδότηση για τα προγράμματα, τα περιβαλλοντικά και τα γεωργικά προτείνει ένα 60%. Ξέρω πως πάρα πολλά κρατημέλη, πάρα πολλές περιφέρειες έχουν προβλήματα με τη συγχρηματοδότηση. Θεωρώ πως όλοι γνωρίζουμε αυτά τα προβλήματα και θα πρότεινα πραγματικά να δημιουργήσουμε οριζόντια μέτρα, αλλά όχι στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης ε, και να μην παρεμβούμε δηλαδή στο ποσοστό συγχρηματοδότησης, γιατί φαίνεται θετικό, αλλά στην πράξη θα σημάνει μείωση για πολλές χώρες που έχουν φιλόδοξα αγροτοπεριβαλλοντικά ε, προγράμματα. Και δεν θέλω ε, βεβαίω να απαλλάξω από τις ευθύνε τους και τους εθνικούς υπεύθυνου, γιατί συχνά υπάρχει η δυνατότητα να μειώσουν το συνολικό όγκο για να εξοικονομήσουν κάποιους εθνικούς πόρους. Αυτό δεν είναι νομίζω σωστό για την συνεργασία καινοτομία και τα λοιπά. Ναι, οπωσδήποτε και την 100% χρηματοδότηση. Θα ήθελα να πω πως δεν είναι αυτό δική μας δουλειά και επιπλέον δεν είναι δική μας δουλειά να υποστηρίζουμε μεγάλες επιχειρήσεις παραγωγής ε, σπόρων. Θα πρέπει και τα μικρά περιφερειακά ε, γεωργικά Ινστιτούτα να έχουν την δυνατότητα να κάνουν την έρευνα αυτή. Η γραφειοκρατία αναφέρθηκε ήδη και κατά την άποψή μου οι προτάσεις ε, του εισηγητή λόγω της πολυπλοκότητας και της καλής θέλησης παρόλα αυτά ε, θα καταλήξουν να είναι δύσκολες στην εφαρμογή τους. Πρέπει λοιπόν εδώ πέρα να καταβάλουμε μια προσπάθεια οι προτάσεις Κομισιόν και του Ισηγητή να απλοποιηθούν για να εφαρμοστούν και στην πράξη. γιατί είναι δυσκολότερο και για τις μικρότερες επιχειρήσεις να χρηματοδοτηθούν έτσι. Και θα χαιρόμουν να έχουμε κάποιες πιο φιλόδοξες ε, προτάσεις Έχουμε αυτή την ευκαιρία και πρέπει να το κάνουμε γιατί αυτό πραγματικά μόνο τους γεωργούς θα ωφελήσει, τους παραγωγούς και την ύπεθρο. Και με τέτοιες προτάσεις πρέπει να πάμε στην διαπραγματεύση. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ Ελίζαβεθ, ο Αντιπρόεδρος Πόλσον και μετά Σμιτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα περιμένω λίγο μέχρι να βρείτε τα ακουστικά για τη γλώσσα ειδικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κάπουλα Σάντος γιατί ήταν εξαιρετική η δουλειά που έκανε και σε διαφορά μέρους υπολείπους εγώ θα έλεγα ότι κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ καλό να προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία εξ αρχής και να επιδιώκουμε το συγκερασμό των ε, διαφόρων όρων ε, απόψεων. Δεν είναι ιδεολογικό το θέμα. Είναι πολύ πιο σημαντικό να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε και μην ξεχνάτε η ισχύσεν τη ενώση για να επιτύχουν και οι προσπάθειές μας. Ε, ε, δεν είναι καταστροφικό, ξέρετε, αυτόματα το να συμφωνήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν πρέπει να διαφωνούμε για να διαφωνούμε. Κάτι άλλο τώρα. Όταν πραγματικά αρχίσουμε την συζήτηση και εξετάζουμε την πραγματικότητα σε όλες τις, τις λεπτομέρειες, ε, μήπως θα έπρεπε όλοι να έχουμε κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι θα πρέπει ε, να λάβουμε δεόντως υπόψη τις νέες προτεραιότητες, ε, τις δημοσιονομικές ε, περικοπές. Όταν μιλάμε κυρίως για τον πυλώνα 2, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι απαραίτητο να παραμείνει για να είναι εύρο στη γεωργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάποιες περικοπές επειδή επιβάλλονται, αλλά όχι με καταστροφικό για τη γεωργία τρόπο τρόπο. Σε σχέση τώρα με τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου, προφανώς ε, τα 30% του πυλώνα 1 πρέπει οπωσδήποτε να είναι μια βασική γραμμή που όλοι θα μπορούν να ακολουθήσουν και σε ένα ορισμένο βαθμό συμφωνώ με τους ε, πρασίνους ε, ότι δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε με τα προαιρετικά συστήματα και να υπάρξει απώλεια του 30% του εισοδήματος ή της ενίσχυσης. Δεν νομίζω ότι αυτός ο τρόπος σκέψης ε, είναι οικολογικός. Ε, δηλαδή σε κάποιο βαθμό θα πρέπει να εφαρμόσουμε την πολλαπλή συμμόρφωση. Σε σχέση με την πράσινη γεωργία υπάρχει ένα ζήτημα που έχει κέρια σημασία ε, δεδομένης της σημερινής κατάστασης. Πρέπει οπωσδήποτε για τις ε, αρρώσιμες σε ε, να επιτρέπουμε να προστατεύονται από το χιόνι και από την βροχή ε, και από τις δύσκολες κλιματικές συνθήκες. Η Γερμανία έχει χρησιμοποιήσει ένα δορυφορικό σύστημα ελέγχου. Εγώ πιστεύω ότι είναι παράξενο να μην ε, χρησιμοποιούμε ε, αυτά τα τεχνολογικά μέσα για να διαπιστώσουμε ποιες ε, εκτάσεις είναι πράσινες και ποιες όχι. Θα καταθέσω σχετική τροπολογία κύριε Σάντος. Πιστεύω ότι πέρα από αυτό υπάρχει άλλη μια λεπτομέρεια για την ύπεθρο για τις περιοχές που βρίσκονται σε δυσμενέστερη κατάσταση. Ποιο είναι αυτό το θέμα λοιπόν πάση θυσία πρέπει να ε, προασπίσουμε την ε, βιοποικιλότητα. Ε, οφείλουμε να προστατεύσουμε την φύση. Και σας μιλώ εδώ για τις διάφορες ε, ποικιλίε φυτών και ράτσες εκτινοτροφικών ζώων. Αυτή η βιοπικιλότητα θα πρέπει να ε, προστατευτεί και να διασφαλιστεί για το μέλλον. Γιατί όλο ένα και περισσότερο ε, ανάγουμε σε κεντρικό επίπεδο όλη τη διαχείριση, αλλά δεν μπορούμε για τους σπόρους να έχουμε μόνο τεράστιες επιχειρήσεις την ε, αγροβιομηχανία και ας μην ξεχνάμε και τα ζώα. Δηλαδή σε τοπικό επίπεδο πρέπει να προφυλαχθούν οι διάφορες ράτσες ζώων και φυτικές ε, ποικιλίε. Ε, δεν είναι επειδή με έχει πιάσει η νοσταλγία αγαπητοί φίλοι. Το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό για τα παιδιά και για τα εγγόνια μας. πρέπει να παραμείνει άθικτη η βιοπικιλότητα γιατί στο μέλλον θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις βασικές παραδοσιακές παραδοσιακές για να αναπτύξουμε καινούργιε. Τέλο, ε, σε όλε αυτές τι συζητήσει, ε, μιλάμε για το πρασίνισμα, για το περιβάλλον, ε, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορούμε να εισάγουμε το πρασίνισμό ως νέο μέρος της ε, νέας υγειονικής ε, πολιτικής. Ε. Αλλά σας παρακαλώ, όσοι είσαστε από την Ήπεθρο, ξέρετε όπως και εγώ ότι σε καμία περίπτωση δεν θα έχουμε βιο... βιώσιμη Ήπεθρο εάν δεν κατοικείται η Ήπεθρο Δηλαδή πρέπει να λειτουργεί και η κοινωνική ζωή

χρειάζεται ένας κοινωνικός ιστός και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να αναπτύξουμε τα χωριά, τους μικρούς οικισμούς, ε, την ύπεθρο και δεν είναι τόσο απλό να θεωρούμε ότι οι νέοι και οι νέες θα παραμείνουν στην ύπεθρο, δηλαδή πρέπει να προβλέψουμε κάτι για αυτόν που θέλει ε, να είναι γεωργός. Ε, πώς θα είναι μια γυναίκα γεωργός, παραδείγματος χάρη, αν δεν υπάρχει βρεφονιπιακός σταθμός, πού θα τα είναι το παιδί. Πρέπει να δείτε και ε, πώς θα λειτουργήσει το κοινωνικό σύστημα στην Ήπεθρο για να φέρουμε την ζωή στην Ήπεθρο, ούτω ώστε να είναι βιώσιμη και η γεωργία. Ευχαριστώ. Αντιπρόεδρε Πόλσον. Σμιτ και μετά Σκότα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ λογικά αυτά που μας είπε η κυρία Πάουλσεν και θα την υποστηρίξω και υποστηρίζοντα ταυτόχρονα έτσι την προσέγγιση του εισηγητή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο με τεχνητό τρόπο πρέπει να διαφοροποιείται η Επιτροπή μας εάν έχουμε την ίδια θέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευτυχή σύμπτωση είναι αυτό και θα πρέπει να είμαστε και ικανοποιημένοι ε, γνωρίζοντας ε, κυρίως πόσο δύσκολες θα είναι οι διαπραγματεύσεις. Καλύτερα να υπάρχει μικρότερη απόσταση ανάμεσα στο και την Επιτροπή από ότι ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, γιατί έχει ασχοληθεί η Επιτροπή ε, με διάφορου ε, φακέλου για την ποιότητα, παραδείγματο χάρη, που δεν ταιριάζουν με την πολιτική τη Λισαβόνα. Χρειαζόμαστε συμμάχου τουλάχιστον ε, για τα δημοσιονομικά θέματα. Οπότε όταν προσωμιάζουν οι προτάσει μα την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγώ δεν θα ανησυχούσα σε σχέση με τι άμεσε πληρωμέ, γιατί εγώ από πλευρά τη ομάδα μου ασχολούμαι με το θέμα τη ανάπτυξη υπαίθρου, αλλά για τι άμεσε πληρωμέ Ήθελα να πω το θέμα της επιλεξιμότητας των μονίμων ευόσκο το ε, δηλαδή τα αγροστόδη που διεγράφησαν ε, ε, μας ικανοποιούν. Ευχαριστούμε για αυτήν την αλλαγή, για την ανάπτυξη της υπέτρου υποστηρίξου σε σχέση με την αναβολή της μεταρρύθμισης για τις περιοχές που βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση. Θα δεχτούμε πολύ μεγάλη πίεση, αν δεν μείνουμε στη θέση μας εάν τα κράτη-μέλη δεν έχουν κάνει επαρκή ε, χαρτογράφηση, δεν έχουμε τα πετούμενα στοιχεία για να προσδιορίσουμε αυτέ τι περιοχέ και να εισαγάγουμε το νέο σύστημα. Κατά τα λοιπά, για τα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα και εμεί είμαστε υπέρ τη ε, ε, μικρότερη δυνατή γραφειοκρατία σε σχέση με τη λήψη απόφαση όταν μιλάμε για την προθεσμία των δύο μηνών. Έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία ω προ τα χρονοδιαγράμματα και θα συμφωνήσουμε για το 30% τώρα για τα αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα και για τις πληρωμές ε, στα πλαίσια του Natura 2000 είμαστε υπέρ. Όπως φαντάζεστε, επίσης ε, χαιρόμαστε που υπάρχουν δυνατότητες ε, για την εμφάνιση της συνεργασίας ανάμεσα στους γεωργούς για τα αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα. Θέλουμε να διευρυνθούν αυτά τα πολύ αποτελεσματικά μέτρα που προτείνεται. Τώρα μια, ένα άλλο διαφορετικό φιλοσοφικό θα έλεγα ζήτημα για την ανταγωνιστικότητα των νέων γεωργών και την πληρωμή των 35.000 ευρώ. Διαφωνούμε κάθετα και δεν πρόκειται να αλλάξουμε γνώμη γιατί δεν επενδύουμε έτσι ε, στο μέλλον ε, της γεωργικής πολιτικής. Είναι μεταμφιεσμένη κοινωνική πολιτική και ε, μη αποδεκτή χρήση των δημοσίων κονδυλίων κατά αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό σας είπα ότι είναι φιλοσοφικό το θέμα, δηλαδή το να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα των γεωργών για αυτές τις επενδύσεις ε, δεν είναι καλή ιδέα γιατί έτσι ω κανίβαλοι θα ε, κατασπαταλήσουμε ε, τα χρήματα του δευτέρου πυλώνα και θα ενισχύσουμε όχι τους γεωργού, ή το πρασίνισμα αλλά τους κερδοσκόπους. Σε σχέση τώρα <coughs> με τη χρήση της άρδευση. Ε, να γνωρίζετε ότι υπάρχει σοβαρή διάσταση απόψε ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Δεν πιστεύουμε πάντω ότι τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα ε, τα προάγουμε όταν με τεχνητό τρόπο τα εισαγάγουμε στο δεύτερο πυλώνα και μιλάμε για την άρδευση ε, των ξηρών αλλά παραγωγικών γεών Ω προ τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου θέλουμε όντως η προσέγγιση να είναι από κάτω προ τα πάνω και τα κράτη-μέλη γνωρίζουν πολύ καλά ποια είναι τα συμφέροντα, ποια είναι τα ε, προβλήματα και ιδιαιτερότητε σε κάθε περιοχή. Και άρα θα πρέπει να έχουν ηγετικό ρόλο κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων Επίσης, ε, προγράμματα συνεργασίας ανάμεσα στους ε, γεωργούς, ε, κοινή διοκτησία γης, χρήση, κοινή χρήση εξοπλισμού. Τέτοια μέτρα θα μας επιτρέψουν να προωθήσουμε την πολιτική ανάπτυξη της υπαίθρου. Θα έχουμε μάλιστα ηγετικό ρόλο και θέλουμε όχι να αποδυναμωθούν, αλλά να εμπλουτιστούν οι σχετικές προτάσεις. Θα συνεργαστούμε μαζί σας για αυτό το φάκελο και σας συγχαίρουμε διότι μέχρι στιγμής έχετε συμπεριλάβει πολλές και διαφορετικές απόψεις. Ευχαριστώ. Τελευταίος ο Τζανκάρλο Σκοτά είναι ο τελευταίος και όδης εισηγητής. Ο Τζανκάρλο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και συνάδελφοι. Εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Θέλω όμως ευθύ αμέσω να σταθώ σε ορισμένα σημεία. Διαβάζοντας τους τελευταίους μήνες την πρόταση της Κομισιόν διαπίστωσα ότι ο όρος γυναίκα δεν αναφέρεται πουθενά. Θα έπρεπε λοιπόν να εισάγουμε τον όρο, πόσο μάλλον στο άρθρο 8, για τα θεματικά υποπρογράμματα. Και στο 20 για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό, ε, έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ε, γυναίκες ε, γεωργούς. Επίσης, πολλές γυναίκες γεωργοί που, έχουν γεωργικές εκμεταλλεύσεις ξεπερνούν τα 60 χρόνια ηλικίας. Πάντα μέσα στο άρθρο 20, παράγραφος 20, όπως αναφέρθηκε από τον συνάδελφο, Πιστεύω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να δημιουργήσουμε ένα ταμείο εγγύσεων για τους νέους γεωργούς, θεωρώντας ότι η βοήθεια για την εγκατάσταση νέων γεωργών αν έρχεται στους 70.000 ευρώ. Η πρόταση της Κομισιόν ε, ήταν, ε, η αντίδραση της Κομισιόν σε αυτή μου την πρόταση ήταν θετική. Για το 2014-2020 θα μπορούσαμε να έχουμε ταμεία εγγύσεων στα πλαίσια του ΦΕΤ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των νέων γεωργών. Είμαι πεπισμένος ε, ότι παρότι έχουμε και επιδοτήσεις ε, και ταμεία, ένα τέτοιο είδος ε, κονδυλίου θα, θα δημιουργούσε κίνητρα στους νέους να εγκατασταθούν στην Γεωργία. Ευχαριστώ Τζαν Κάρλο. 20 συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Θα έλεγα λοιπόν ότι από τώρα και στο εξή θα έπρεπε να έχουμε τρία λεπτά ο καθένας. Ο Μισελ Νταντά και μετά ο Ζωζέ Μποβέ. Ο Μισελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από σήμερα, νωρίς από σήμερα το πρωί ξεκινήσαμε να μιλάμε και μιλήσαμε για πράσινες ενισχύσεις, για περιβάλλον. Εγώ θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η γεωργική δραστηριότητα είναι καταρχόν οικονομική δραστηριότητα. Είμαστε λοιπόν εδώ για την προάσπιση ενός οικονομικού κλάδου που διατρέφει 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους, που εξάγει και συμβάλλει στον πλούτο της Ευρώπης και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Πίσω από αυτήν την οικονομία κρύβονται άντρες και γυναίκες και τα μέτρα τα οποία θα λάβουμε πρέπει να τους επιτρέψουν καταρχήν να συνεχίσουν να ζουν. Άκουσα τις παρατηρήσεις του Πολωνού συναδέλφου, τις καταλαβαίνω. Αλλά υποχρεούμε να του πω ότι σε ορισμένες χώρες της παλαιάς Ευρώπης μία γρήγορη μείωση της υποστήριξης θα οδηγήσει στην πλήρη εξαφάνιση των γεωργικών εκμετελεύσεων. κυρίως στην κτηνοτροφία που θα δεχτεί τις μεγαλύτερες επιπτώσεις και αν δεν μπορέσουμε εμείς να διατηρήσουμε αυτές τις ενισχύσεις σε ορισμένες περιφέρειες, η γεωργία αυτών των περιφερειών θα εξαφανιστεί. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τις προτάσεις που υπέβαλε. Εγώ θα ήθελα να το ρωτήσω δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, για το greening, το πρασίνισμα. Εμένα το πρασίνισμα καταρχήν δεν μου δημιουργεί πρόβλημα. Η ενίσχυση του πρασινίσματος θα πρέπει να αποσυνδεθεί από τη βασική από τη βασική ενίσχυση. Τώρα, το greening πώς το μετράμε, αναεκμετάλλευση ή αναχώρα. Διότι άμα το μετρήσουμε αναχώρα και το μοιράσουμε μετά σωστά, δίκαια στους γεωργούς, θα αποτελέσει ένα σκαλοπάτι. Πρέπει λοιπόν να λάβει θέση το Κοινοβούλιο. Πώς υπολογίζουμε εμεί το πρασίνισμα. Για το νερό. Εγώ σημείωσα ότι θέλατε να κρατηθεί το σύστημα άρδευσης εκεί όπου το νερό αποτελεί τροχοπέδι στην ανάπτυξη της παραγωγής. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί στον δεύτερο να διατηρούμε την οδηγία πλαίσιο για το νερό ενώ εμείς στην Επιτροπή Γεωργίας είχαμε πει ότι θα έπρεπε να βγάλουμε αυτή την οδηγία πλαίσιο όταν αυτή δεν εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Για τις ζώνες με φυσικές δυσκολίες το να συμπεριλάβουμε τα, τις ορεινές περιοχές δεν ξέρω γιατί όταν μιλάμε εμείς ε, για ζώνες με δυσκολίες, με καταναγκασμούς, με δεσμεύσεις, είναι περιοχές οι οποίες ε, έχουν οικολογικές ε, προσταγές να ακολουθήσουν. Τώρα για τα βουνά δεν νομίζω ότι όλες οι περιοχές είναι έτσι. Τώρα, ή ιστορικά στις χώρες μας και με τους μόνιμους βοσκοπο... και οι μόνιμοι βοσκότοποι, οι λεγόμενοι μόνιμοι βοσκότοποι, καλλιεργούντουσαν πάντα. Δηλαδή κάθε 15-20 χρόνια στην Ευρώπη γυρνούσαμε την, κοργόναμε τις, ε, ε, του, τους βοσκοτόπους για να τους ε, ε να τους ξανακαλλιεργήσουμε ως βοσκοτόπους. Αν δεν υπάρχει αυτό το γύρισμα της γης, αν δεν γίνει αυτό το όργωμα, τότε χάνεται η δυναμική ε, και η ποιότητα των ε, όπως επίσης και οι τυφλοπόντικες αυξάνονται Ευχαριστώ. Να δούμε πώς θα διαχειριστούμε το χρόνο στη διάθεσή μας. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ρολόι. Δύο μισή λεπτά ο καθένας, γιατί αλλιώς δεν τελειώνουμε. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν εγώ να κάνω μία εισαγωγή. Αυτή τη βδομάδα θα ξεκινάει η διάσκεψη του Ρίο και έχω την αίσθηση ότι γυρνάμε, γυρίζουμε την πλάτη σε αυτές τις ε, δια, διεθνείς ανησυχίες που εκφράζονται και τα σχέδια τα οποία επεξεργαζόμεθα εμείς ή αντιφάσκουν πλήρως με τους στόχους, τους παγκόσμιους στόχους. Η κυρία Μαγίνες πολύ σωστά είπε ότι χρειάζεται προπολογισμό. Για να υπάρξει προπολογισμό χρειάζεται μια συμβατή πολιτική. Για να έχουμε συμβατή πολιτική θα πρέπει να ε, οι πολίτες ε, να δεχθούν να τους φορολογήσουμε για να χρηματοδοτήσουμε αυτή την πολιτική. Με διάφορα στοιχεία που έχουμε σήμερα σε αυτή την έκθεση εμείς απομακρυνόμεθα από την νομιμότητα, διότι απομακρυνόμεθα και από τη συνάφεια των στόχων μας. Σύντομα, δεν θέλω να σταθώ στα θετικά, γιατί όπως είπαμε δεν μιλάμε για τα τρένα τα οποία φτάνουν στην ώρα τους, μιλάμε για αυτά που καθυστερούν, δηλαδή για τα αρνητικά. Το τα πρώτα αρνητικά. Για τις μικρές εκμεταλλεύσεις, εγώ πιστεύω ότι έχουμε ένα προχώρημα, γιατί μιλάμε για μία έλαφρή μικρή αύξηση, 1500 αντί 1000 ευρώ. Υπάρχει όμως και κάτι το επικίνδυνο ότι αυτές οι μικρές εκμεταλλεύσεις στο τέλος της εκμετάλλευσης θα είναι 35.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό στο τέλος της ε, αλυσίδας της διαδικασίας φτάνουμε στις 35.000 ευρώ, πράγμα το οποίο δεν επιτρέπει για μια αξιοπρεπή σύνταξη, για τις ενισχύσεις. Υπάρχουν αντιφάσεις μέσα στο κείμενο. Εφόσον εμείς έχουμε μία προοδευτική μείωση η οποία δεν βελτιώνεται στην πραγματικότητα διότι η διαδικασία λέει ότι από το 70 και το 80% 100 περνάμε αντί να έχουμε μία οροφοποίηση φτάνουμε σε οροφές των ε, 150 αντί των 120 ευρώ. Αυτό το οποίο όμως είναι επικίνδυνο είναι η παράγραφος που λέει ότι η εκμετάλλευση ε, όταν γίνεται εταιρικά ε, ξεφεύγει από αυτήν την οροφή. Στο πρώτο κείμενο το είχαμε στα γαλλικά και το βρίσκω πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Ανοίγουμε εμείς ορίζοντα εδώ για τις εταιρείες, ε, δεν υπάρχει πλαφόν για το πρασίνισμα της ΚΑΠ θα είναι κρίμα. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και την ε, κυκλωτικότητα των ε, καλλιεργιών ε, στην, μέσα στη διαδικασία του πρασινίσματος. Μείωση των, οικολογικών, των γεών οικολογικού ενδιαφέροντος κατά 2% δεν μου φαίνεται καλό. Εξαίρεση από τα μέτρα πρασινίσματος. Επιστήνω την προσοχή σας ότι είναι επικίνδυνο να βάζουμε μέσα ειδικέ περιβαλλοντολογικές ε, ε, σημάνσεις διότι αυτές οι σημάνσεις μπορεί να είναι και αποτέλεσμα λόμπι. Ε, νομίζω ότι θα έπρεπε να τα βγάλουμε λοιπόν. Τώρα για το θέμα των ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών ήδη εξηγήθηκε αλλά μεταξύ των Γιωργών πιστεύω ότι είναι ενδιαφέρον να προσέξουμε. Δημιουργούμε μία επικίνδυνη κατάσταση και δεν είναι νορμάλ να λέμε από τη μια θέλουμε να ερχόμαστε στα ίδια δικαιώματα. Λοιπόν, μία φορά μιλάμε για την, ΠΑΚ, για το βρίσκω απαράδεκτο να αντιδρούμε έτσι. Συνεχίζω. Είναι θέμα οργάνωσης των συζητήσεων. Εγώ θεωρώ αξιοθρύνητο για ένα θέμα τόσο σημαντικό να μην έχουμε μία χρήσιμη συζήτηση με τον απαραίτητο χρόνο. Δεσμεύουμε τη Γεωργία για έξι χρόνια. Τελειώνω με αυτό το στοιχείο. Δεν είναι νορμάλ. Θεωρώ επικίνδυνο σε ένα από αυτά τα άρθρα να λέμε ότι μία χώρα μπορεί να περιορίζει κάτω από το 30% το 2014. Έχω κι άλλα να πω, αλλά θα τα πω γραπτός. Η συζήτηση όμως σήμερα δεν γίνεται ούτε σοβαρά, ούτε με τρόπο επαρκή. Κυρίε και κύριοι, αν συνεχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε πριν τι 12.30. Παρακαλώ, δύο λεπτά έκαστος και έκαστη. Ας μην επαναλαμβάνουμε αυτά που ήδη έχουν ακουστεί και μπορείτε εξάλλου να υποβάλλετε και γραπτός παρατηρήσει. Δύο λεπτά παρακαλώ καθένας, γιατί αλλιώ δεν θα προλάβουμε. Χωρί μικρόφωνο. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το οποίο ανέλαβε <clears throat> και κυρίως να συνδυάσει όλες τις οπτικές. Άλλοι θα το βρίσκουν πολύ φιλόδοξο, άλλοι λιγότερο, άλλοι συνάδελφοι πολύ πράσινο, άλλοι λιγότερο πράσινο. Ο στόχος αυτής της Επιτροπής είναι να μπορέσουμε να έχουμε μια στεναρή θέση ως Κοινοβούλιο για να αμυνθούμε των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Ε, ευχαριστώ που λάβατε υπόψη την ευελιξία για το greening. Και αυτό δηλαδή για να μπορέσουμε να συνδεθούμε με την ουσία της ευρωπαϊκής ε, γεωργίας. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από ότι εγκαταλελειμμένη ύπεθρος. Πρέπει λοιπόν αυτά για τα μέτρα για το πρασίνισμα να είναι μέτρα υλοποίησιμα για τους, για τους γεωργούς μας ή και να είναι ουσιαστικά. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Κάπουλας να αποκλείσει τους συνεταιρισμούς, διότι δεν θα ήταν κατανοητό από τη μια να, προκαλούμε εμεί τους γεωργούς μας να ενώνονται, να οργανώνονται κτλ και από την άλλη μεριά να πλήττουμε τις, ε, τους συνεταιρισμούς. Θεωρώ ότι είναι καλό να διευρύνουμε τη μεταβατική περίοδο για να προσαρμοστούμε στη νέα βασική πληρωμή για τις χώρες οι οποίες έχουμε ιστορικά δικαιώματα θα έπρεπε ίσως ε, να προσαρμοστούμε κάπως περισσότερο για να μην έχουμε απότομες αλλαγές ε, μεταξύ των παραγωγών μας. Σύμφωνο απόλυτα με την ανάγκη να ενσωματώσουμε το στοιχείο το, του προβληματισμού της γυναίκας μέσα στην ε, πολιτική της υπαίθρου, όχι γιατί δηλαδή οι γεωργοί μας θα πρέπει να τις παντρευτούν, αλλά για οι γυναίκες να μπορέσουν να πάρουν μεγαλύτερο, να αναλάβουν μεγαλύτερο ρόλο στην ζωή της υπαίθρου. Πρέπει να έχουμε μία καλύτερη τοποθέτηση για ορισμένα θέματα, αλλά θα πρέπει να έχουμε και μία στεναρή θέση ως κοινοβούλιο για να εγγυθούμε το μέλλον των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και πάλι θα ήθελα αρχίζοντας να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Σίγουρα ήταν ε, λέει η κυρία Ντότσο, «Ε, πάρα πολύ δύσκολο και περίπλοκο το ζήτημα και χρειάστηκε να αντιπεξέλθει σε μεγάλες δυσκολίε. Α αρχίσω με τα δημοσιονομικά θέματα. Σήμερα συζητάμε για ε, προτάσεις χωρίς να γνωρίζουμε την πρικοδότηση των δύο πυλώνων. Ε, αναμένονται βεβαίω περικοπέ και ω εκ τούτου θεωρώ ότι θα έπρεπε να εστιάσουμε την προσοχή μας ε, ε, στο να καταλάβουμε που, σε ποια σημεία μπορούμε να στηρίξουμε αποτελεσματικά τη γεωργία και τους γεωργούς. Επίσης θα πρέπει να μειώσουμε το γραφειοκρατικό ε, και δεν καταλαβαίνω πώ θα το επιτύχουμε αυτό ακολουθώντα είτε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε την έκθεση του κυρίου Σάντους. Γίνουν πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα και δεν ξέρω πρέπει να συνεχίσουμε την εξέταση όλων αυτών των ζητημάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, επιδιώκει να ελέγχουμε και να διοικούμε τα πάντα από τις ευρυξέλλες. Είναι πολύ πιο λογικό να αφήσουμε πολλά πράγματα στα κράτη-μέλη. Υποστηρίζω την ευελιξία ε, σε επίπεδο κράτους μέλους ε, και περιφέρειες και δεν θα υποστηρίξουμε σε καμία περίπτωση τις απόπειρες που γίνονται ούτω ώστε να παρεμβαίνουν οι Βρυξέλλες για το πώς καλλιεργούμε στα 27 κράτη-μέλη με όλες ε, τις εναλλακτικές ε, λύσεις ε, που μπορούν να υπάρξουν για τόσο διαφορετικές καταστάσεις. Σε σχέση με τη μεταφορά των πονδυλίων από τον ένα πυλώνα στο άλλο ήταν πάρα πολύ λεπτό το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ όμως δεν ασχολούμαι με αυτό. Θα ήθελα να ασχοληθώ με τη δική μου εκλογική περιφέρεια στη Βόρεια Ιρλανδία. Γιατί να κατευθυνθούμε προς ένα ε, καταποκοπή ποσό για το πρασίνισμα. Μία τέτοια εφάπαξη πληρωμή ε, θα έχουμε πολύ σοβαρές επιπτώσεις στον τομέα των εγωπροβάτων και της εκτροφής ε, των ε, βοηδών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνυπολογίσουμε αυτούς τους παράγοντες ε, και οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη γνώμη μου θα ε, θέσουν σε κίνδυνο στον τομέα των βοητών και των αγοπροβάτων τη ζωή ε, και την επιβίωση των εκμεταλλεύσεων. Θα έπρεπε τουλάχιστον να επιδιώξουμε μια επταετή περίοδο σύγκλησης. Ως προς το πρασίνισμα του πρώτου πυλώνα και πάλι, παρά είναι περιοριστικό, πάλι οι Βρυξέλλες προσπαθούν να βρουν μια ενιαία λύση για όλους. Δεν λειτουργούν αυτά τα πράγματα Χρειαζόμαστε ευελιξία, χρειαζόμαστε αυτό τον κατάλογο, το μενού και τη δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε ε, στις ε, τοπικές ιδιαιτερότητες ως προς ε, τις καλλιεργητικές πρακτικές, το κλίμα και το καθεξής. Για τις περιφέρειες, ποιος μπορεί να συμμορφωθεί με όλες τις απαιτήσεις σε περιφερειακό επίπεδο κατά 95% η Ιρλανδία είναι βοσκότοπη. Υπερβαίνουμε τους ορισμούς που Μύχη. Mm. Ε, ορίζονται. Οπότε ε, ε, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τα μέτρα αυτά που προτείνονται για τις περιοχές που υπερβαίνουν κάποια ποσοστά. Ζητώ συγγνώμη και θα σταματήσω τώρα απλώς. Πραγματικά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια <coughs> σε σχέση με αυτό που μας προτείνει ο εισηγητής για τους παραδοσιακούς λιμόνες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε επίσης ιδιαίτερα με την παραγωγή τροφίμων και την έννοια του ενεργούς γεωργού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Ντότς, Καρινιέτα και Ντόφμαν τώρα παρακαλώ. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī vēlos pievienoties visiem tiem, kas apsveic mūsu kolēģi Kapulašu Sānu. Ευχαριστώ, θα υποστηρίξω και εγώ όλους αυτούς που συνεχάρισαν τον εισηγητή. Όντως εργάστηκε με εξαιρετικό τρόπο. είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, για τους ε, Λετονούς ε, γεωργούς να ρυθμίσουμε όλα αυτά τα αισθήματα που αποσχολούν εξάλλου τους γεωργούς όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα καταθέσω σχετικές τροπολογίες. Η βασική προτεραιότητα για μας είναι οι άμεσες πληρωμές που θα είναι ομοιόμορφες ε, σε όλα τα κράτη-μέλη. Η τροπολογία 9 είναι πολύ θετικό βήμα, αλλά βάσει αυτού Ακόμη και το 2020 οι άμεσες πληρωμές στη Λετωνία θα είναι κατά 2,5 ε, φορές χαμηλότερες σε σχέση με ε, πληρωμές που γίνονται σε άλλα κράτη-μέλη, άρα δεν θα ισχύουν ε, ε, ίσοι όροι ανταγωνισμού ε, και ανοίγουμε το παράθυρο για διαφθορά. Όταν ισχυρίζονται κάποιοι ότι θα πρέπει να συνδυάσουμε τις πληρωμές και τα ποσοστά των πληρωμών με το γενικότερο μέσο όρο. Ας δούμε ποια είναι η κατάσταση στις βαλτικές χώρες προς το παρόν. Η Λετωνία λαμβάνει το 30% μόνο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Για να επιτύχουμε λοιπόν ίσως όρους ανταγωνισμού, ε, χρειαζόμαστε αλλαγή της ε, κλίδας κατανομής ε, για να πλησιάσουμε το ποσοστό του 0,66% ε, ούτως ώστε να μην υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Προτάθηκε επίσης μία τριετή περίοδος σύγκληση. Όμως εγώ θεωρώ πως στις περιοχές όπου οι πληρωμές είναι τόσο χαμηλές όσο στις βαλτικές χώρες ε, χρειαζόμαστε αλλαγές ε, ήδη από την πρώτη χρονιά, δηλαδή το 2014. Δεν ζητούμε γενεοδορία, δεν ζητούμε θυσίες ε, από κανέναν όπως το έθεσαν κάποιοι συνάδελφοι. Οι γεωργοί των χωρών ε, της ε, Βαλτικής. Ε, δεν περιμένω από αυτούς που παίρνουν τριπλάσια ενίσχυση από την Ευρώπη να θυσιαστούν. Όχι, δεν ζητάμε αυτό απλώς. Διεκδικούμε δικαιότερους όρους ανταγωνισμού Και μην ξεχνάτε πώς ε, ξεπούλησαν τις βαλτικές χώρες της Σοβιετική Ένωση οι δυτικές ε, χώρες ε, στο παρελθόν. Αυτές οι νέες χώρες έχουν την ίδια άποψη όλες και θα πρέπει να ακουστεί και η φωνή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ να είστε λίγο πιο σύντομοι στι μελλοντικέ σας παρεμβάσει, Ευχαριστώ, ελπίζω να προλάβω. Ευχαριστώ για τον εισηγητή για τη δουλειά που έχει κάνει. Δύο-τρία πράγματα θέλω να αναφέρω. Στα ζητήματα ενεργός Γεωργός Μικρή Γεωργή πρέπει να προσέξουμε πόση επικουρικότητα υπάρχει. Αν αφήσουμε πολλές επιλογές στα κράτη-μέλη, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε αυτή την κατάσταση την οποία έχουμε σήμερα με τις μειονεκτικές περιοχές. Δηλαδή να διαφέρει η κατάσταση τελείως από κάθε κράτος μέλος. Για τον πρώτο πυλώνα τώρα. Η πρόταση του εισηγητή είναι να γίνει πιο να επιβραδυνθεί η σύγκληση μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό είναι λάθος, θεωρώ, πως, ε, όπως είπε και η κυρία Καλινιέτε, θα πρέπει ε, ό,τι είπαμε για τη σύγκληση μεταξύ των κρατών μελών να ισχύει και για τη σύγκληση Εντό των κρατών μελών και εκεί πέρα είναι πιο σοβαρά τα πράγματα. Π.χ. στον τομέα του γάλακτος υπάρχουν οι γεωργοί οι οποίοι παράγουν γάλα και λαμβάνουν 10 φορές περισσότερες άμεσες ενισχύσεις από τον πρώτο πυλώνα από άλλους γαλακτοπαραγωγούς. Δεν μπορεί κάποιος να μου πει πως δεν είναι αυτό στρέβλωση της αγοράς εντός της ίδιας χώρας. Η αδικία αυτή πρέπει να σταματήσει και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν και θεωρώ πως αυτό το οποίο πρότεινε η Κομισιόν 7 ε, χρόνια δηλαδή ε, νομίζω πως έχει αποδειχθεί στη Γερμανία πως μπορεί να ισχύσει και χωρίς μεγάλες ε, ανατροπές. Δύο παρατηρήσεις ακόμα για το δεύτερο πυλώνα μειονεκτικές περιοχές Θεωρώ πως υπήρξε μία έκθεση πέρσι, την οποία ούτως ή άλλως ψηφίσαμε, μία σχετική έκθεση και αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε. Κάτι άλλο δεν αναφέρθηκε. Για τα ειδικά πριν, για τις τοπικές ομάδες δράσης που προτείνει η Κομισιόν για πολύ έτσι ωραία ε, έργα στο πλαίσιο του LEADER Κάποιος ήταν μεθυσμένος μάλλον όταν τα έλεγε αυτά. Η Κομισιόν εδώ πέρα μοιράζει πριμ και λεφτά. Δεν είναι λογικά πράγματα. Ξεπέρασα το χρόνο, νομίζω, κατά μισό λεπτό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν είναι εδώ. Μα δεν σας κατάλαβα κύριε Πρόεδρε, όπου εγώ δεν άκουσα το όνομά μου πουθενά. Λοιπόν, μη μου αφαιρέσετε καιρό, ε, ε χρόνο. Ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι τις γνώμες ορισμένων συναδέλφων σαν αυτή του κυρίου Λάιον ότι πρέπει να είναι πιο τολμηρή η πρόταση. Διότι εμείς σήμερα συζητάμε για τις εφαρμοστικές λεπτομέρειες χωρίς όμως να συζητούμε τους στόχους για τη μετα... της μεταρρύθμισης. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Καπόουλας διότι έκανε μια πολύ σημαντική προσπάθεια για, την... για να υπάρχει μια συλλογική συνένεση. Βέβαια τα ιστορικά δικαιώματα βλέπουμε ότι θα εξαφανιστούν, αλλά παρόλα αυτά τον ευχαριστώ. Επίσης από το κάπινγκ θεωρώ πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι βγάλαμε τους συνεταιρισμούς. Δεν μπορούμε εμείς να επιβαρύνουμε τους γιοργούς... οι οποίοι είναι οργανωμένοι. Τον ευχαριστώ που ενσωμάτωσε επίσης το κοινωνικό κριτήριο διότι προσδίδει μεγαλύτερη ηρεμία στα κράτη-μέλη όταν πρέπει αυτά να εφαρμόσουν τα μέτρα αυτά. Για το greening εγώ έχω ιδιαίτερες ανησυχίες. Καθιστά πιο ευέλικτο το greening ο εισηγητής. Αναφέρ, ξεχνάει όμως τον οικολογικό ρόλο ορισμένων καλλιεργών όπως είναι τα, καλλιεργιών όπως είναι τα όσπρια. Όπως επίσης ξεχνάει και το καπνό. Καλλιέργειες που είναι πολύ σημαντικές για τη χώρα μου. Εγώ πιστεύω ότι ο εισηγητής θα πρέπει να ορίσει τι εστί ως ιστορική καλλιέργεια. Επίσης, εγώ δεν είμαι ικανοποιημένη με τον όρο μόνιμος βοσκότοπος, διότι έτσι αγνοεί βασικούς οικολογικούς ε, τόπους, ε, όπως ας πούμε στην Ισπανία ή ε, η Ντέσα που είναι τεράστιες εκτάσεις με οικολογικό ενδιαφέρον. Πρέπει να έχουμε έναν ορισμό πολύ πιο ακριβή όπου θα εκπράζονται σαφώς όλες οι, όλοι οι φυσικοί, όλες οι φυσικού ενδιαφέροντος περιοχές στην Ευρώπη. Πολύ σωστά βέβαια είπανε πολύ ότι θα πρέπει να εκλεπτύνουμε όλα αυτά τα κριτήρια για τη χορήγηση των ενισχύσεων όπως είπε και η κυρία Κώστιγκερ ότι τα λεφτά πρέπει να τα παίρνουν πραγματικά αυτοί οι οποίοι δουλεύουν τη γη. Γιατί τη μεταφορά τώρα από το δεύτερο στον πρώτο πυλώνα. Ή όλοι ή τίποτα. Για τους Γιοργούς υπάρχει ένα θέμα πολύ σοβαρό το οποίο δεν λάβαμε υπόψη. Η οι νέοι γεωργοί, παραγωγοί που κληρονομούν εκμεταλλεύσεις οι οποίες ήδη είναι εταιρείε και επιβαρύνονται και επιβαρύνονται ιδιαίτερα κατά την το πέρασμα της κληρονομιάς. Γιατί αν έχουμε ας πούμε τρία αδέρφια δεν θα έχουν ποτέ το 50% της εταιρεία. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ βεβαίως. Ε, θέλουμε να ξαναμιλήσει ακόμα ο εισηγητής ε, και η Κομισιόν. Κυρία Ματία, λοιπόν. ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον συνάδελφο Κάπουλας αλλά θα ήθελα να πω κάτι για τον greening. Το θεωρώ λίγο φιλόδοξο για την εφαρμογή κάτω από τα 5 εκτάρια και θα ήθελα επίσης να προσθέσουμε στην αναφορά που έγινε για τα φρούτα και τα σπεριδοειδή. Για το κάπινγκ, εγώ υποστηρίζω την πρόταση της Κομισιόν και δεν συμφωνώ με τη μείωση των κατοφλίων του συγητή. Θέλω όμως σύγκριση για τις άμεσες πληρωμές στα κράτη-μέλη και είμαι απόλυτα ε, κατά της τοπικής καινοτόμου συνεργασίας. Αυτό το μέτρο, όπως είπε και ο κύριος Ντόρφμαν, απλώς καλύπτει μερικούς που θέλουν να μοιράσουν κονδύλια. Θέλω να ρωτήσω όμως την Κομισιόν και να επιστήσω την προσοχή του εισηγητή. Για τους ιστορικούς βοσκότοπους. Εγώ μίλησα για permanent grassland, μόνιμους βοσκότοπους στην εκθεσή μου. Εδώ μιλάμε για ιστορικούς βοσκότοπους. Είναι θέμα ορολογίας που θα πρέπει να ομοιομορφοποιήσουμε μεταξύ των εκθέσεων. Διότι έχω την αίσθηση ότι αναφερόμαστε στα ίδια πράγματα. Διότι αναφερόμαστε σε βοσκοτόπους αμφότεροι, όπου έχουμε όμως και, ε, και δέντρα και δεντροκαλλιέργειες. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρχει μία ομοιογενοποίηση της ορολογίας. Είναι απαραίτητη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, νομίζω πως όλοι ε, συμφωνούμε πως θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον ε, εισηγητή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν κατάλαβα το όνομά μου λέει η κυρία Γέγλε. Εν πάση περιπτώσει. Πρώτα απ' όλα οφείλω να ευχαριστήσω τον συγητή. Δεύτερον, το δικό μας ε, σκιώδη συγητή, την κυρία Κέστιγκερ δηλαδή, για το θέμα του δεύτερου πυλώνα. Εκεί προσυπογράφω 100% όσα είπε η κυρία Κέστιγκερ. Κατόπιν, θα ήθελα να μάθω από τον συγητή ποιοι είναι οι λυποί γεωργοί. Τι εννοείται. Τι εννοείται με ιστορικούς ιστορικές χορτολιβαδικές εκτάσεις. Μετά, τρίτον, το leader, όπως το είχαμε μέχρι τώρα, την προσέγγιση που είχε. Οι πολίτες επιτόπου αποφασίζουν ποιο έργο θέλουν να κάνουν. Αυτό νομίζω πως είναι η σωστή προσέγγιση και για το μέλλον. Αυτό το οποίο προτείνει η Κομισιόν είναι λάθος από πάνω προς τα κάτω. Και τέλος γνωρίζω πως οι γυναίκες ε, συμπεριλαμβάνονται εδώ πέρα ρητός από ό,τι γνωρίζω. Απλά είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω στην Υπεθρό, ρητός σε ορισμένα σημεία να μιλήσουμε για τις γυναίκες και την ισότητά τους στο πλαίσιο των προγραμμάτων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρόδους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Εγώ τώρα διαφωνώ κάπως. Θεωρώ πως η έκθεση της Κομισιόν είναι καλή ως βάση εργασίας και ακόμη καλύτερο είναι το, ε, οι βελτιώσεις οποίες επέφερε εδώ πέρα ο συνάδελφος. Οι συνάδελφοι λένε να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Έχουμε τα 58 δισεκατομμύρια ως αφετηρία σήμερα και πρέπει νομίζω σοβαρά να δείξουμε πως θέλουμε ένα πρασίνισμα και στηρίζουμε την Ευρώπη 2020. Εάν λοιπόν ε, κάνουμε το λεγόμενο greenwashing έτσι για τα μάτια μόνο πρασίνισμα δεν θα είναι σωστό. Μην ξεχνάμε πως ε, πρέπει να φροντίσουμε να βρούμε και απήχηση και στο Κοινοβούλιο εκτός της Επιτροπής μας, της Επιτροπής μας. Τώρα, για το πλαφόν. Είμαι εναντίον, δεν νομίζω πως θα είναι σωστό. Είχαμε ήδη μία ψηφοφορία και ήταν σαφές, νομίζω, 75% των συναδέλφων θεωρούν πως πρέπει να υπάρξει κάποιο πλαφόν. Οπότε, τι να κάνουμε, πρέπει να το συνδιαμορφώσουμε Επίσης για συνεταιρισμούς και τα λοιπά όπου συνεταιρίζονται πολύ μικροί γεωργοί πρέπει να ληφθούν υπόψη και καλά το κάνατε. Ενεργός γεωργός, ε, καλά τα είπε ο Λουίς, λέει θέλουμε να έχουμε με έναν αρνητικό κατάλογο να ορίζουμε το τι δεν είναι. Αυτό νομίζω είναι το σωστό. Ε, μείωση της γραφειοκρατίας, ναι. Εδώ πέρα Βεβαίω, για ποιον χτυπάει η καμπάνα, χτυπάει για το εθνικό κράτο. έλεγχο του ελέγχου δεν χρειάζεται. Και βεβαίω για το πρασίνισμα. Πρέπει να πρασινίσει ο πρώτο πυλώνας. Ο δεύτερο πυλώνα υπάρχουν ήδη όλα αυτά και να πούμε ξεκάθαρα στου υπόλοιπου βουλευτέ, πώ είμαστε διατεθειμένοι να μεταρρυθμίσουμε τι άμεσε πληρωμές. Εάν δεν το κάνουμε αυτό δεν θα έχουμε πλειοψηφία. Γι' αυτό είμαι υπέρ του πρασινίσματος και είμαι πεπισμένη πως με καλή βούληση θα τα καταφέρουμε να έχουμε και αυτό το 7% περιοχών οικονο... Ε, ε, οικολογικής προτεραιότητας. Και ίσως έπρεπε νομίζω να επικεντρωθούμε στο επίπεδο της περιφέρειας. Θεωρώ λοιπόν πως το πρασίνισμα να γίνει από τα 10 εκτάρια και πάνω. Οτιδήποτε άλλο είναι αντιπαραγωγικό γιατί έχουμε πολλές εκμεταλλεύσεις στην Ευρώπη που είναι πάρα πολύ μικρές. Και δεν είναι δυνατόν ένα κομμάτι της Ευρώπης να πρασινίσει και ένα άλλο όχι. Γι' αυτό ζητάω εγώ να το ορίσουμε στα 10 εκτάρια. Ναι, βεβαίω πρέπει να αποκτούν οι διπλές πληρωμές για το ίδιο πράγμα και να υπάρχει ο δεύτερος πυλώνας όπως τον περιέγραψε η κυρία Πάλουσεν για να εφαρμοστεί. Συνοψίζοντας, θεωρώ πως δεν πρέπει να κάνουμε πρασίνισμα για τα μάτια μόνο. Γιατί θεωρούμε πως έτσι θα ε, ικανοποιήσουμε τους γεωργούς. Εγώ είμαι πεπισμένη πως μπορούμε να τα εξηγήσουμε αυτά στους ε, γεωργούς και θα μας πιστέψουν αν ε, εξηγήσουμε και τα της χρηματοδότησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Φάινμαν και μετά Αντές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω πια, αλλά δεν πειράζει. Οι Τσέχοι Γεωργοί είναι κατά τον, του μέτρου αυτού του πρασινίσματος για λόγους αρχής. Γιατί για λόγους ιστορικούς στη χώρα μας έχουμε το μεγαλύτερο μέγεθος γεωργικής εκμετάλλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τη Σλοβακία και μου ζήτησαν οι Σλοβάκοι Γεωργοί να πω το ίδιο πράγμα. Τι θέλω να πω λοιπόν, είμαι κατά αυτής της αρχής του πλαφών γενικώ και άρα είμαι κατά της ε, πρότασης ε, του εισηγητού για να γίνει πιο περιοριστική η πρόταση αυτή σε σύγκριση με αυτά τα οποία προτείνει η Κομισιόν. Να σας ρωτήσω επίσης ε, τι εννοείται με, την, ε, με τον αποκλεισμό των συνεταιρισμών. Γιατί στο κείμενο που έχω μπροστά μου στα τσεχικά δεν ξέρω εάν ισχύει το πλαφόν για τους ε, συνεταιρισμούς. Καλό θα ήταν λοιπόν να έχουμε μία νομοθεσία και όχι μία να υπερισχύει της ε, άλλης. Επίσης να πω σύντομα κάτι για τους νέους αγρότες και το... την πάυση ε, γεωργικής δραστηριότητας. Νομίζω πως έχει σωστά διατυπωθεί. Επίσης η ηλικία των 65 ετών ανταποκρίνεται στην ηλικία συνταξιοδότησης και στη γύρανση του πληθυσμού και καθιστά δυνατόν ε, το να δοθεί η εκμετάλλευση σε επόμενες γενιές. Επίσης υποστηρίζω αυτό το οποίο είπε η κυρία Καλνιέτε όταν μίλησε για δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη στην κατανομή των πληρωμών σε όλους τους γεωργούς, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω πως πρέπει να δούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μία αγορά όπου ανταγωνίζονται οι γεωργοί μεταξύ τους και θα ήταν λάθος να υπάρχουν παρεκκλήσεις και διαφορές ε, μεταξύ κρατών μελών. Μιλάω για τις ε, πληρωμές αυτές. Οπότε στηρίζω όλες τις προτάσεις που ακολουθούν αυτό το δρόμο και τελικά ελπίζω να ξεφορτωθούμε όλες αυτές τις διαφορές. Σας ευχαριστώ. <coughs> να πω κάτι για τους συνεταιρισμούς. Στα νέα κράτη-μέλη έχουμε διαφόρων ειδών συνεταιρισμούς. Γι' αυτό από τους ορισμούς μπορείτε να βγάλετε συμπέρασμα για, το, για ποιον ακριβώς συνεταιρισμό πρόκειται. Ο κύριος Ντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον ε, κύριο Κάπουλας ε, Σάντος για τη σκληρή δουλειά που έχει κάνει και να κάνει. Αν ε, τώρα λέμε κάποια πράγματα, στόχος δεν είναι η κριτική, θέλουμε όλοι να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις προτάσεις σου. Και θέλω και εγώ να συμφωνήσω και με όσους ευχαρίστησαν και, τα, και τους και τη Μαρία Μαγκίνες αλλά και τον ε, George Λάιον ε, και τον κύριο Νίκολσον και τον κύριο Ντόρφμαν και με αυτούς συμφωνώ, οπότε δεν θα τα επαναλάβω τα όσα είπαν. Θεωρώ πως πρέπει να προσπαθήσουμε το πρασίνισμα αυτό να είναι πιο λογικό και πιο κοντινό στην πράξη και πιο ευέλικτο στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό θεωρώ, Λουίς, πως πρέπει να δούμε το θέμα του μενού, το οποίο αποφασίσαμε με 90%. Μην ξεχνάμε αυτό το οποίο είπαν οι συνάδελφοι. Εάν υπάρχουν περιφέρειες που υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο 20% δεν χρειάζεται να εφαρμοστεί τίποτα άλλο. Πρέπει να δούμε λοιπόν το επίπεδο της περιφέρειας, αλλά δεν είναι κοντά νομίζω στην ε, πράξη το να έχουμε κάπου ένα 20% και μετά να αφαιρείται άλλο ένα 7% ή 14% από την παραγωγή. Επίση πρέπει να συζητήσουμε την ε, πρότασή σου για μεταφορά των αδιάθετων κονδυλίων του πρασινίσματος στον δεύτερο πυλώνα. Δεν ε, το θεωρώ αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό. Ίσως θα ήταν καλύτερο να πάνε αυτά ως ε, αύξηση της βασικής ενίσχυσης. Αυτά και τελειώνω εδώ πέρα για να μην υπερβώ το χρόνο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, κύριε Κάπουλα Σάντος, σας ευχαριστούμε για την έκθεση. Απλοποίηση και μείωση γραφειοκρατίας πάντα τα αναζητούμε, αλλά εδώ πέρα πρέπει να είναι μαθηματική η γεωργία για να βγάλουν κάποια άκρη. Άρα εγώ δεν βλέπω καμία απλοποίηση. Επίσης δεν υπάρχει εδώ πέρα διαπραγματευτικό περιθώριο είναι τσίμα τσίμα τα πράγματα. Δύο-τρία πράγματα τώρα. Οι περιοχέ οικολογική προτεραιότητα, ο εισηγητή εδώ πέρα συμπεριλαμβάνει κάποια νέα πράγματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πω πρέπει να υπάρξει ένας ε, νέο υπολογισμό ε, των ε, επιλέξιμων περιοχών. Στη Γερμανία, παραδείγματο χάρη, κάποιε εκτάσει εξαιρούνται, τα είπαμε όλα αυτά ήδη πολλέ φορές υπάρχει αγρανάπαυση, κάθε δρόμος ο οποίος υπάρχει επίσης ε, θεωρείται ότι δεν χρησιμοποιείται και επίσης ε, σε συνεργασία δύο αγροτών ε, να υπολογιστούν αυτές οι περιοχές. Ναι, είναι λογικό, θα οδηγήσει νομίζω και σε περισσότερες συνεργασίες. Και ε, βεβαίως ε, θα δούμε το τι μπορεί να γίνει συνολικά σε μια περιφέρεια. Τώρα για παραδοσιακούς, ε, παραδοσιακές χορτολιβαδικές εκτάσεις ετέθη το ζήτημα. Μειονεκτικές περιοχές νομίζω πρέπει να παραμείνουμε στην απόφαση πως ε, θα πρέπει να μείνουμε στο 2015 για νέα πρόταση της Κομισιόν. Αλλά δεν θα πρέπει να προδικάσουμε τίποτα και να πούμε στην Κομισιόν πρέπει να δει τα βιοφυσικά κριτήρια, όχι αν είναι απλά, να αφήσουμε ανοιχτό το τι πρόταση θα κάνει η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Χάρτιν. Χάρκιν και Έντουαρτς. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τον εισηγητή, διότι εργάστηκε πολύ σκληρά για αυτό το θέμα. Πολλοί μίλησαν για το μεγάλο ελέφαντα <laughs> μέσα στο δωμάτιο, δηλαδή το ζήτημα που κανεί δεν θέλει να συζητήσει, αλλά που είναι το σημαντικότερο, δηλαδή ο προπολογισμό πρέπει να επανερχίσουμε τι προτεραιότητε μα. Κάποιε παρατηρήσει προ τον εισηγητή. Πρώτον, ω προ την ανακατανομή των αμέσων πληρωμών χρειαζόμαστε μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο και σίγουρα ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση ο γιατί αναγνωρίζει το θέμα του περιορισμού των απολειών ε, και ε, δεν μπορούμε όμως να περιοριστούμε σε αυτό. Χρειαζόμαστε ισορροπία, όπω είπε και ο Τζιμ Νίκολσον. Ε, μιλάμε συνέχεια για μικροκαλλιεργητές και θέλει να ασχοληθούμε και με τι μεγάλε εκμεταλλεύσεις. Μα χρειαζόμαστε ισορροπία γιατί και οι δύο συμβάλλουν στη βιωσιμότητα τη υπαίθρου και με τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία τη Ιρλανδίας επιβεβαιώνονται οι ανησυχίε σε σχέση με τα βοηθή και τα εγωπρόβατα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην υπάρξει μεγάλη απώλεια λόγω των αλλαγών. Για το, τα χρόνια της ενεργοποίηση. Συμφωνώ με τον εισηγητή, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό από το 2009 ως το 2011. Κάθε χρόνο πρέπει να ξέρουμε με σαφήνεια ότι ε, με μονομένο τρόπο μπορεί να επιδιώξει κανείς την ενεργοποίηση. Για το 70% τώρα των ε, οικολογικών περιοχών ε, ε, θα πρέπει να συνδέσουμε αυτό το μέτρο με ένα νέο ορισμό ε, ε, των χωρών οικολογικής εστίασης για τη δέσμευση αζότου παραδείγματος χάρη. Όπως είπαν δε και άλλοι συνάδελφοι, για το πρασίνισμα χρειαζόμαστε ένα πραγματικό μενού τώρα ε, για την... Ε, ε, θα θέλαμε κι εμείς τα κράτη-μέλη να έχουν διακριτική ευχαίρεια ώστε να ορίσουν τα κριτήρια στη συνέχεια τώρα για τις πληρωμές προς τους παλιούς γεωργούς. Στην χώρα μου το, η κατάσταση έχει ως εξής. Είναι, υπάρχει μεγάλη κατάτμιση και σίγουρα θα είναι θετικό το μέτρο για την Ιρλανδία. Ο ενεργός γεωργός είναι πολύ καλύτερη η δική σας ε, πρόταση, γιατί λαμβάνει υπόψη ε, ε, οικονομικά κριτήρια και άλλα που θα εξασφαλίσουν ότι θα λαμβάνουν ενεργή γεωργή τις πληρωμές τώρα σε σχέση με τα κριτήρια θα πρέπει να δούμε αν έχουμε επαρκή και αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για τον προσδιορισμό ε, των γεωγραφικών ζωνών ω προ τη βιωσιμότητα. Συμφωνώ με τον εισηγητή, δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε μόνο στα περιβαλλοντικά μέτρα. Χρειαζόμαστε ολιστική προσέγγιση, ούτω ώστε τα οικονομικά, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα τη γεωργία να συνδυαστούν και άρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το ρόλο των γυναικών από αυτή την άποψη. Συμφωνώ και με τη Μαρίτα Πάουλσεν πρέπει να είμαστε ρεαλιστές ω προ τι προτάσει Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και ε, να προστατεύσουμε την βιοποικιλότητα. Τέλος, ε, χρειαζόμαστε μια προσέγγιση από κάτω προ τα πάνω και σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει κοινοτική καθοδήγηση για την εφαρμογή των μέτρων. Σας ευχαριστούμε. Έλγο τώρα. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή γιατί προσπαθεί να επιτύχει μια εξισορροπημένη θέση και είναι ιδιαίτερα δυσχερή η κατάσταση. Ε, η νομιμοποίηση, η αποτελεσματικότητα των κατευθυντηρίων γραμμών είναι με ένα από τα βασικότερα προσκόμματα. Έχει εργαστεί με εξαιρετικό τρόπο. Επίση, δεν γνωρίζουμε τον προπολογισμό και με αυτό ω δεδομένο είναι σχεδόν αδύνατο να αποφασίσουμε για τι περικοπέ και τι ανακατανομέ των κονδυλίων. Για το πρασίνισμα ε, προβλέπω να ανακύπτουν διάφορα ε, προβλήματα και άρα χρειαζόμαστε ένα κατάλογο εναλλακτικών λύσεων, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία. Αυτή η ενιαία λύση για όλου ε, δεν μπορεί να αποτελέσει την πιο πρόσφορη μέθοδο για όλα τα κράτη-μέλη και θέλει ο εισηγητή να μειώσει κατά 30% τη απόλυση εισοδήματο για του γεωργού. Δεν νομίζω ότι είναι επαρκέ αυτό. Με αυτό το 30% που προτείνει ο εισηγητή γνωρίζω ότι ένα μεγάλο αριθμό γεωργών Λοιπόν, ε, θα ε, πληγούν από μικρή απώλεια εισοδήματος. Ε, θα πρότεινα το 10% αλλά θα Αναγνωρίζω ότι χρειάζεται σκληρή δουλειά για να το επιτύχουμε. Για την καταποκοπή πληρωμή μέχρι το 2019 νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δυσεφάρμοστη αυτή η λύση και πρέπει να επανεξεταστεί. Για τον ορισμό του ενεργού, του ενεργού γεωργού ε, κοιτάξτε, ο ενεργό γεωργό είναι ραχοκοκαλιά και τη γεωργία και τη ε, αγροβιομηχανία ε, και πιστεύω ότι οι προτάσει αυτέ μπορούν να έχουν σοβαρέ ε, παρενέργειε για, πλέον, για του πλέον παραγωγικού τομεί τη γεωργία. Θα πληγεί και η βιομηχανία ω αποτέλεσμα εφαρμογή αυτών των μέτρων. Αν τελικά εγκριθούν, να καλωσορίζω την απόφαση να αναβληθεί η επανεξέταση των ε, περιοχών που βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση. Νομίζω ότι ήδη έχουν επομιστεί ένα υπερβολικό ε, άχθος ε, κατά κεφάλι και χρειάζονται σοβαρότατε και σκληρέ διαπραγματεύσει για να αλλάξουμε ε, την κατάσταση για το ε, καθεστώ συνταξιοδότηση ε, των μικροκαλλιεργητών και την καταποκοπή πληρωμή. Επιτρέπονται οι επενδύσει πλέον στο κεφάλαιο και στον εξοπλισμό και τελικά η μεταφορά των δικαιωμάτων πληρωμών από τον ένα γεωργό στον άλλον θα έχει αρνητικά αποτελέσματα κυρίως για τους μικρολιεργητές, για τους νέους γεωργούς, τροπολογία 28 και τους νέους γεωργούς που θα δίνουν ε, τις εγγυήσεις ε, για την ε, βιώσιμη γεωργία. Είναι λογική η πρόταση και θα μπορούσε να είχε θετικά αποτελέσματα. Όμως θα πρέπει να επανεξετάσουμε διεξοδικότερα τον, όλο τον μηχανισμό. Ε, βρίσκω ενδιαφέρουσα την πρόταση συγχρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα που καταθέτει ο εισηγητής ε, και δεδομένων των δημοσιονομικών περιορισμών που γνωρίζουν κάποια κράτη-μέλη. Νομίζω ότι αυτό θα αποτελούσε λύση για τη συγχρηματοδότηση, όμως ε, θεωρώ ότι χρειάζονται σαφείς και αυστηροί κανόνες σε σχέση με το τι είναι αποδεκτό, δηλαδή ιδιωτική συγχρηματοδότηση σε όλη αυτή την αλυσίδα πρέπει να επανεξεταστεί προτού εισαθεί στην νομοθεσία. Και τέλος, Πρόεδρε, θα θέλω και πάλι να αναφερθώ στην απλούστευση, ε, διότι στην αρχή της συζήτηση μας απασχόλησε αρκετά αυτό το θέμα και μείωση της γραφειοκρατίας. Δεν ε, βλέπω πώς θα μπορούσαμε να το επιτύχουμε αυτό με τα μέτρα που προτείνονται. Ε, ένα μενού εναλλακτικών λύσεων σίγουρα θα μας βοηθήσει ως προς τις επιθεωρήσεις και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, αλλά τέλος πάντων έχουμε τώρα ξεκινήσει πλέον ένα πολύ μια πολύ σοβαρή συζήτηση που θα παρακολουθήσουμε εκ του και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Νικολέ... Κυρία ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ, Έχω. Πρόεδρε. Ε, έχασα την αρχή της συζήτησης, αλλά επειδή πίσω κάθεται ένας ε, ε, φοβερός Ολλανδός δημοσιογράφος, θα παρακολούθησα όλα μέσω του Twitter. Ε, ε, θα ήθελα για το πρασίνισμα να πω κάποια πράγματα, γιατί από ό,τι κατάλαβα απασχόλησε πολλούς από τους συναδέλφους. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να έχουμε το μενού με τις αναλλακτικές λύσεις και τους υπολείπους που είναι κατά. Ε, πιστεύω ότι το μεγαλύτερο τμήμα της πολιτική μου ομάδα είναι σε αυξημένου πρασινίσματο με βιοποικιλότητα, ανανεώσιμε πηγές ενέργειας, καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, αποτελεσματική χρήση των πόρων, νέε επενδύσει κτλ. Ε, αλλά και τώρα στρέφομαι προς τους ε, πράσινου. Αν δώσετε στα κράτη-μέλη αυξημένη ευελιξία, θα <laughs> πρέπει από την άλλη πλευρά και αυτό το εργαλείο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να καλύψουμε το χάσμα μεταξύ των δύο ε, στρατοπέδων. Αν αυξήσετε λοιπόν την ευελιξία, δηλαδή αυτό που ζητούν ε, οι υπουργοί να μα δώσουν τα λεφτά και μετά θα αποφασίσουμε τι θα τα κάνουμε, δεν πιστεύω ότι θα λειτουργήσει το σύστημα. Είμαι ε, βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άρα θα πρέπει να καταλήξω σε μια ευρωπαϊκή λύση. Αν δώσουμε ευελιξία, λοιπόν θα είναι και πρέπει να είναι και πιο υπόλογα τα κράτη-μέλη. Παραδείγματο χάρη, τα κράτη-μέλη να μπορούν να πάρουν τέσσερι από τι έξι εναλλακτικέ λύσει, αλλά θα, πρέπει να καταδείξουν σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιοι είναι οι στόχοι που θα επιτευχθούν τα επόμενα έτη δεδομένη τη κατάσταση και δεδομένη μια βασική γραμμή ελαχίστων δηλαδή πραγμάτων που θα πρέπει να επιτύχουν. Δεν θέλω να είναι πιο φιλόδοξα τα κράτη-μέλη, αλλά οι φιλοδοξίε αυτέ πρέπει να είναι ρεαλιστικέ και το μενού πρασινοποίηση για την Ολλανδία προ το παρόν ναι, δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Να το δείξετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς, τι θέλετε να επιτύχετε, πώ θα το επιτύχετε και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει και κριτήρια και να σα κρίνει μετά ναι, την εκπνοή μια συγκεκριμένη συγκεκριμένη σε περίοδο. Οπότε ένα είδο σύμβαση που θα χρησιμοποιείται κατά τη γνώμη μου ε, και στα διαρθρωτικά ταμεία. Λοιπόν, έτσι μπορούμε να καλύψουμε το χάσμα ανάμεσα σε αυτού ε, που είναι υπέρ του μενού και αυτών που είναι κατά. Όχι να αυξήσουμε την ευελίξια, αλλά είπα να είναι και η λογοδοσία ε, αυξημένη για τα κράτη-μέλη και θα ήθελα να ακούσω και την άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι εγώ είμαι ρεαλίθρια πολιτική άποψη για να δω πώ τι πολιτικέ ομάδε είναι υπέρ του μενού και εδώ πώ οι υπουργοί είναι υπέρ αυτού του μενού των εναλλακτικών λύσεων, προς τα εκεί κατευθυνόμαστε. Ε, οπότε παρακαλώ να μας βοηθήσετε και απευθύνομαι τώρα και στους πράσινους και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτύχουμε λοιπόν να έχουμε μεγαλύτερη λογοδοσία γιατί αλλιώς ε, θα φτάσουμε μπροστά σε ένα τείχο. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Και εγώ με τη σειρά μου τον εισηγητή. Γιατί κατάφερε να συνδυάσει όλες τις απόψεις που ακούστηκαν κατά τη συζήτηση. Εγώ λοιπόν κοιτάζω, έχω δίπλα μου και το, την έκθεση αλλά και το κείμενο της Κομισιόν. Η Κομισιόν λέει ότι τα κράτη που δέχονται άμεσες πληρωμές θα πρέπει να τις περιορίσουν κατά το 1 τρίτο. Ο εισηγητής όμως με τη σειρά του λέει οι χώρες εκείνες που βρίσκονται κάτω από το 70% του κοινοτικού μέσου όρου θα πρέπει να μειώσουν κατά 30%. Εγώ δεν βλέπω εδώ όμως καμία διαφορά. 30% είναι 30% είναι το 1 τρίτο ούτε παραπάνω ούτε λιγότερο. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν τη διαφορά μεταξύ της πρότασης ε, της Κομισιόν και της πρότασης του εισηγητή, διότι αυτό το οποίο λέει η έκθεση δεν λέει τίποτα. Συμφωνώ με την αρχή της σύγκρισης, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να επεξεργαστούμε καλύτερα τα εκατοστία ποσοστά. Επίσης ανησυχώ και για το θέμα του μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που είναι πολύ άριθμες ε, στη Ρουμανία. Εγώ πιστεύω ότι η ΚΑΠ, η νέα ΚΑΠ δεν θα είναι καθόλου απλό να, εφαρμοστεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κάπουλα Σάντα ε, γιατί ήταν πολύ δυσκερέ το έργο και τα κατάφερε παρόλα αυτά ε, πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα λοιπόν ε, να σχολιάσω κάποια μέρου στοιχεία για το πρασίνισμα. Καλό είναι για του γεωργού να έχουν πολλέ εναλλακτικέ λύσει. Θέλω όμω, όπω ο κύριο Ντελάν, ότι για να, είναι, ε, για να έχουν νόημα αυτά που κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να αυξήσουμε και την ευελιξία και την λογοδοσία. Ε, αυτό είναι το, η μόνη λογική λύση. Ε, τα, οι παραδοσιακοί λιμόνες θα πρέπει να προσδιορίσουμε αυτήν την ε, έννοια. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αν δεν ε, γνωρίζουμε τι ε, υπογράφουμε, τι δεχόμαστε, γιατί αυτό επηρεάζει και την στήριξη, την ενίσχυση και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε αν δούμε ιστορικά τι έχει γίνει. Άρθρο 9, το αρχικό κείμενο. για οι τροπολογίες δεν λένε τίποτα για, τις, ε, για τους ε, κλιματολογικούς περιορισμούς σε σχέση με τον ε, αριθμό των καλλιεργειών. Μιλάνε μόνο για το εμβαδό των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθούμε στους φυσικούς ε, περιορισμούς, διότι σε κάποιες χώρες όταν έχει κάποιος λίγο πάνω από 20 εκτάρια, δεν μπορεί κανείς να περιμένει, ε, όντας ρεαλιστής, να έχει διαφορετι... τρεις διαφορετικές καλλιέργειες ε, ο Γεωργός ε, σε αυτή την έκταση. Για τους ε, νέους Γεωργούς, πιστεύω ότι στα κράτη-μέλη που έχουν τις ενισχύσεις στο δεύτερο πυλώνα για τους νέους γεωργούς, και για τα κράτη που θέλουν να υπερβούν την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, λοιπόν, πιστεύω ότι το σύστημα θα πρέπει να είναι προαιρετικό. Ευχαριστώ. Θέλω να ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και παρεμπιπτόντως έχω και εγώ ένα ζήτημα που θέλω να σχολιάσω για τις μεταβατικές περιοχές, ε, δηλαδή που βρίσκονται στο 75% ε, του μέσου ορού του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, στις ε, μητροπολιτικές περιοχές ισχύει μια διαφορετική πραγματικότητα σε σχέση με την Ήπεθρο και οπωσδήποτε θα πρέπει να συνυπολογιστεί αυτό διότι δεν θέλουμε να περιορίσουμε το φάσμα των εναλλακτικών λύσεων των ε, περιοχών της Υπέθρου που έχουν σημειώσει μεγαλύτερη ανάπτυξη σε σχέση με άλλες. Αυτά από πλευρά, μου και τώρα θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Πατσίσκου για τις άμεσες πληρωμές πρώτα απ' όλα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Κάπουλα Σάντος ε, για την εξαιρετική του έκθεση, πολύ αναλυτική, ε, προβληματισμένη και σε βάθος. Εγώ Πιστεύω ότι για το θέμα του ορισμού των βοσκοτόπων μπορούμε να συνεργαστούμε για να βρούμε έναν κοινό ορισμό αποδεκτό. Πρέπει επίσης να πω ότι ήδη η Κομισιόν ε, ε, δέχθηκε έναν πιο πλατή ορισμό που να συμπεριλαμβάνει τους παραδοσιακούς βοσκοτόπους όπως η Ιντεέζα στην Ισπανία ή το Μοντάδο στην Πορτογαλία ή το σύστημα των βοσκοτόπων που έχουμε στη Σκοτία ή στην Σουηδία. Για τα άλλα σημεία θα ήθελα να πω ότι στην έκθεση του κυρίου Κάπουλα Σάντος υπάρχουν προτάσεις για το κάπινγκ, θα τις εξετάσουμε. Θέλω όμως επίσης να πω ότι για τον ορισμό του ενεργού Γιώργου... Ε, στην έκθεση του υπάρχει υποχρεωτικότητα ε, ως όρος. Εγώ θα ήθελα να κρατημέλη να ορίσουν αυτά τα κριτήρια και, αν είναι μετά θα είναι υποχρεωτικά. Για τη σύγκληση μεταξύ κρατών μελών αναγνωρίζω ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα, αλλά εγώ δεν μπορώ παρά να σημειώσω τις προτάσεις του κυρίου Κάπουλα Σάντος και τις ε, τοποθετήσεις των άλλων, ε, συναδελ... Ε, των άλλων μελών αυτής της Επιτροπής, διότι είναι κάτι το οποίο διαπραγματευόμαστε μέσα στα πλαίσια του πολιτούς δημοσιονομικού σχεδίου. Τώρα, για τη σύγκληση μέσα στο κράτος μέλος μεταξύ γεωργών, αυτό το οποίο διαπιστώνω είναι ότι στην έκθεση του κυρίου Κάπουλα Σάντος Υπάρχει ένας ε, ρυθμός σύγκλησης ε, που θα μπορούσε να, να είναι, ο οποίος είναι πιο περιορισμένος από αυτό το οποίο προτείνουμε εμείς. Θα ήθελα επίσης πολύ σύντομα να σταθώ στην ευελιξία μεταξύ πυλώνων. Ε, πρέπει να κρατήσουμε σημαντικά ποσά στον πρώτο πυλώνα κατά τρόπο ώστε μέτρα όπως το πρασίνισμα να βρουν τη θέση τους. Επίσης εκφράζουμε ανησυχίες για τις διατάξεις εκείνες ε, οι οποίες θα μας επέτρεπαν να αλλάξουμε με τις μεταφορές κάθε χρόνο, να αλλάζουμε τις μεταφορές κάθε χρόνο, γιατί αυτό θα επιβάρυνε την ανάπτυξη της υπαίθρου. Τώρα θα να σταθώ λίγο στο θέμα του πρασινίσματος, είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και για τις προτάσεις μας και για την έκθεση. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι διαφωνούμε με, διαφωνούμε με μια περιορισμένη προσέγγιση του θέματος. πολύ το, αποδυναμωμένη προσέγγιση, πολλοί το ζήτησαν σε αυτή την Επιτροπή. Αν ακολουθήσουμε όμως εμείς αυτήν την προσέγγιση δεν θα έχουμε κανέναν τρόπο να, έχουμε, να εγγυθούμε μία ίση και μη διακριτική μεταχείριση μεταξύ των γεωργών των κρατών μελών και των περιφερειών επίσης. Δεν θα είχαμε επίσης τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε ένα άλλο μέτρο το οποίο επίσης υποστηρίζουμε, δηλαδή η ισοδυναμία μεταξύ γεωργικο-περιβαλλοντολογικών μέτρων και greening. Δηλαδή ε, δεν θα μπορούσαν να ε, εφαρμόσουν το greening τα κράτη-μέλη άμα δεχόντουσαν μια πιο περιορισμένη ε, εμβέλεια. Για το θέμα της προαιρετικότητας, ε, χθες έκανα τα σχόλιά μου στην έκθεση Λαβία. Ε, βλέπω ότι είστε ευθυγραμμισμένοι όσον αφορά στην θέση σας. Ε, είστε συνεπείς στις θέσεις σας. Ε, αλλά και εγώ είμαι επίσης συνεπής στις θέσεις μου και λέω ότι δεν συμφωνώ στην προαιρετικότητα. Μπορούμε να δεχθούμε να έχουμε ένα μίνιμουμ εκτάσεων κάτω από το όριο των οποίων δεν μπορεί να εφαρμοστεί για γεωπονικούς λόγους το greening, είμαστε σύμφωνοι. Μπορούμε επίσης να υποστηρίξουμε, να έχουμε ειδική μεταχείριση για, τους, για ομάδες γεωργών σε περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος, τους όρους πρέπει να τους ορίσουμε Επίσης, θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν επαρκείς δικαιολογίες για να έχουμε ένα όριο εκτάσεων ε, που θα επιτρέπουν την εξαίρεση του γεωργού στην οικολογική περιοχή. Εγώ θεωρώ ότι όποια, εμείς θεωρούμε ότι όποια και να, όποιο και να είναι η έκταση όλοι μπορούν κάλλιστα να συμμετέχουν σε αυτές τις περιοχές αυτά για τις άμενες πληρωμές. Τώρα, ε, για την ανάπτυξη της υπαίθρου θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Γέτσικ Πλέβα για να σταθεί στη δεύτερη έκθεση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να εκφράσω τις ευχαριστίες της ε, Κομισιόν στον τον κύριο Κάπουλα Σάντος, για τη δουλειά που έχει κάνει για το σχέδιο έκθεσης για τις άμεσες πληρωμές. Η Κομισιόν θεωρεί πως ε, έχουμε εδώ πέρα μια καλή αφετηρία για την τελική συζήτηση, δείχνει πως αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και επίσης τη λογική πίσω από την πρόταση της Κομισιόν. Προφανώς το έγγραφο προτείνει κάποιες αλλαγές και θα ήθελα σύντομα να αναφερθώ σε κάποιες από αυτές. Να ξεκινήσω με μία από τις τροπολογίες που αφορά τους στόχους ε, της ε, πολιτικής ε, αυτής, συγκεκριμένα το σκεπτικό πως όχι μόνο η Γεωργία αλλά και η νοσοκομεία πρέπει να αναφέρεται ρητός στους στόχους της ανταγωνιστικότητας. Η Κομισιόν αναγνωρίζει πως ο τομέας αυτός συνεισφέρει σε μια ισορροπημένη ανάπτυξη των περιοχών αυτών της Ευρώπης και αυτό αντικατοπτρίζεται νομίζω στο σχέδιο κανονισμού. Εντός των, ε, των ε, περιοχών ε, προτεραιότητας. Άρα θεωρούν πως ο τομέας δασοκομείας ε, νομίζω καλύπτεται επαρκώς από τις προτάσεις της Κομισιόν. Είναι όμως γεγονός πως η Κομισιόν σκοπεύει να μην αναφέρει ρητό στην δασοκομεία στους τρεις βασικούς στόχους της πολιτικής γιατί η συνθήκη δεν μας δίνει κάποια νομική έντολη για πολιτική δασοκομεία στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Χαιρόμαστε για το ότι η Επιτροπή Γεωργίας αναζητά τρόπους να σιγουρευτεί για το ότι θα αντιμετωπίσουμε τις ε, περιβαλλοντικές προκλήσεις του παράδοσης και του μέλλοντος. Το σχέδιο έκθεσης άρα προτείνει το 30% του φακέλου του ΕΤΠΑ του κάθε κράτους μέλους να πάει σε αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Αντί για το 25, η Κομισιόν θεωρεί πως δεν είναι αναγκαίο να γίνουν αυτά νομική απέτηση. Γιατί το βασικό εργαλείο θα είναι η διαδικασία του στρατηγικού προγραμματισμού. Μετά το 2013 τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης θα βασίζονται πολύ περισσότερο στα αποτελέσματα και λιγότερο στις δαπάνες. Ένα άλλο περιβαλλοντικό ζήτημα το οποίο αναφέρει ο εισηγητής είναι η άρδευση και πρέπει πράγματι να βελτιωθεί το κείμενο αυτό που έχουμε τώρα ειδικά η διάκριση μεταξύ νέων και παλιών κρατών μελών. Η Κομισιόν θέλει να το κάνει αυτό στο επίπεδο και συγκεκριμένων νομικών διατάξεων αλλά και παράξεων κατεξιοδότηση. Τώρα θα ήθελα να θέσω κάποια σημαντικά ζητήματα, σημαντικά για την Κομισιόν, όσον αφορά κάποιους φυσικούς ε, περιορισμούς που έχουμε. Η Κομισιόν δεν μπορεί να συμφωνήσει με το σχέδιο έκθεσης του Κοινοβουλίου στο θέμα των ε, περιοχών που έχουν φυσικούς περιορισμούς, περιορισμούς από τη φύση. Το Συμβούλιο αποφάσισε ήδη το 2005 να αλλάξει τους στόχους και τις παραμέτρους του μέτρου. Δεν βλέπουμε λοιπόν, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς μπορούμε να αντιληφθούμε, να καθυστερήσουμε την ε, κοινή μέθοδο ακόμη μία φορά. Επίσης δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί θα πρέπει να υπάρξει ένα ενδιάμεσο σύστημα που θα βασίζεται σε δύο κριτήρια που θα ορίσουν τα κράτη-μέλη και μετά να προτείνουμε ένα σύστημα βιοφυσικών κριτηρίων που θα εφαρμοστεί μετά το 2015. Θεωρούμε πως η προσέγγιση αυτή δεν λύνει το πρόβλημα της διάκρισης μεταξύ των αγροτών που προκαλείται από τα διαφορετικά συστήματα καθορισμού που υπάρχουν. Η Κομισιόν δεν βλέπει το όφελος στο να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν κάποιες αλλαγές οι οποίε θα ισχύσουν για λίγα χρόνια και μετά από λίγα χρόνια ξανά άλλε αλλαγέ. Uh, um, Τώρα θέλω να σχολιάσω το ζήτημα του υψηλότερου ποσοστού συγχρηματοδότησης. Εμείς ε, συζητήσαμε το ποσοστό του maximum ποστού συγχρηματοδότησης για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα του κλίματος. Βεβαίως, μπορούμε να δικαιολογήσουμε το υψηλότερο ποστό για διάφορα μέτρα. Η Κομισιόν ε, επέλεξε διάφορα μέτρα με κάποιο σκεπτικό. Παραδείγματο χάρη θεωρούμε πως η μεταφορά γνώσης είναι θεμελιώδης για μια αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής ε, ανάπτυξης υπέθρου συνολικά. Και πιστεύουμε πως πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των μέτρων που θα έχουν υψηλότερο ποσοστό χρηματοδότησης. Αυτό για λόγους απλότητας, αλλά και γιατί η αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης μπορεί να οδηγήσει τελικά σε μείωση της συνολικής χρηματοδότησης για, για τα συγκεκριμένα μέτρα. Τέλος, το ζήτημα του προγράμματος Leader. Η προσέγγιση που ισχύει για το Leader θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα διαρθρωτικά ταμεία. Στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περίοδου. Αυτό είναι ήδη ένα σημάδι επιτυχίας. Για το λόγο αυτό, το leader βρίσκεται υπό τον κανονισμό των κοινών διατάξεων όλων των διαρθρωτικών ταμείων. Η βασική αρχή του leader είναι η αρχή από κάτω προς τα πάνω, που όπως αναφέρει και ήδη πολλές φορές σήμερα. Δεν αμφισβητείτε. Και οι τοπικές ομάδες δράσης θα παραμείνουν υπεύθυνε για την ανάπτυξη ε, τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών. Κύριε Πρόεδρε, λίγα πράγματα ανέφερα, αλλά ελπίζω να σας ε, έπεισα πως η Κομισιόν παίρνει πολύ στα σοβαρά το έργο της Επιτροπής σας όσον αφορά την πολιτική ανάπτυξη της υπαίθρου και βεβαίως ε, αναμένουμε τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Φαίνεται ότι λαμβάνεται σοβαρή υπόψη τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Γεωργίας. Χαιρόμαστε που είναι τόσο καρποφόρα η συνεργασία μας και οδηγεί σε αυτά αποτελέσματα. Σας ακούσουμε τον εισηγητή μας ε, τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από τη σημερινή συζήτηση και σας ευχαριστώ όλους για την επικοδομητική σας προσέγγιση. Φυσικά δέχομαι τις επικρίσεις και θα ε, προσπαθήσω να καλύψω τις ανησυχίες σας Υπάρχουν κάποια ζητήματα που κατά τη γνώμη μου χρήζουν απλώ και μόνο διευκρίνηση. Παραδείγματο χάρη για την ανακατανομή των κονδυλίων και για να απαντήσω στον συνάδελφο Νικολέσκου. δεν είπε ε, ότι η πρόταση που κάνω εγώ για την ανακατανομή είναι η ίδια με αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ισχύει αυτό. Προτείνει σύγκληση για το 90% του ε, μέσου όρου, ενώ εγώ προτείνω 100% του μέσου όρου και για την ε, Ρουμανία αυτό σημαίνει 400.000 ευρώ για την ε, τωρινή περίοδο προγραμματισμού. Η διαφορά δηλαδή ανάμεσα στις δύο προτάσεις της Επιτροπής και τη δική μου σημαίνει αύξηση του κονδυλίου ε, του πρώτου πυλώνα κατά 400.000 ευρώ. Διαπιστώνεται λοιπόν ε, ότι είναι πάρα πολύ διαφορετικές αυτές οι προτάσεις. Και αυτό θα απαντήσω σε όλους όσους θεωρούν ότι ε, ακολουθώ κατά πόδας την Επιτροπή στις ε, προτάσεις μου. Δεν ισχύει αυτό. Ε, έχουμε ουσιαστικότατες ε, διαφορές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να ευστήσω την προσοχή σα σε ένα άλλο ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο ζήτημα. Αυτό της απλούστευσης. θα ήθελα να καλέσω τους συναδέλφους να διαβάσουν την έκθεσή μου για να βρουν ένα μέτρο που τους φαίνεται πιο περίπλοκο από τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. εγώ αντίστοιχα θα μπορούσα μπορούσα ε, να σα δώσω πολλά παραδείγματα προτάσεων που είναι πολύ απλούστερε από αυτέ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Όταν εγώ προτείνω ότι οι τρει ε, προτάσει του πρασινίσματο ε, θα είναι εφαρμοστε μόνο στις σε πάνω από τα 20 εκτάρια, αποκλείω ανάμεσα στο 70 ε, το 70% και το 80% των γεωργών από αυτήν την γραφειοκρατική υποχρέωση. Υπάρχει ένα ολόκληρο φάσμα προτάσεων σημαντική ε, απλούστευση, όπω παραδείγματο χάρη τα περί ε, δραστηριότητα και αναδιάρθρωση των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Αντί για πέντε ετήσιε πληρωμέ, προτείνω μία πληρωμή, οπότε πέντε γραφειοκρατικέ διαδοχικέ ασκήσει καταργούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να επιβαρύνεται ο γεωργός. Αυτή η πρόταση που κάνω σίγουρα συνεπάγεται πολύ μικρότερη γραφειοκρατία σε σχέση με το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι προφανές ότι υπάρχουν αμφιλεγόμενα ζητήματα ε, και ε, παρατήρησα ότι οι συνάδελφοι που συμφωνούν με την πρότασή μου για την πάυση της δραστηριότητας ε, έχουν παρανοήσει κάποια ζητήματα. Εγώ δεν θέλω να τονώσω την εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας. Το αντίθετο προτείνω οι γεωργοί που είναι 65 χρονών, δηλαδή η νόμιμη ηλικία συνταξιοδότηση, να έχουν ένα επιπλέον κίνητρο για να αποσυρθούν και να ε, ε, ε, επιτρέψουν την εγκατάσταση ενός νέου γεωργού ούτως ώστε να τροφοδοτήσουμε την αναζωογόνηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, διότι σε πάρα πολλά κράτη-μέλη υπάρχουν μικρού μεγέθους εκμετάλλευσης και δεν ε, πιστεύω ότι αν δεν εφαρμοστεί αυτή η πρόταση θα έχει ευνοϊκότερους όρους λειτουργία σε μια μικρή νέα γεωργική εκμετάλλευση διότι το ζητούμενο είναι η οικονομική βιωσιμότητα σε Ζητώ λοιπόν αναδιάρθρωση που θα προσδιορίζουν τα κράτη-μέλη Γι' αυτό τον λόγο προτείνω προαιρετικό σύστημα, διότι αναγνωρίζω ότι για κάποια κράτη-μέλη και για ιστορικούς λόγους η δομή των εκμεταλλεύσεων δεν επιτρέπει την εφαρμογή του συστήματος και γι' αυτό προτείνω να είναι υποχρεωτικό το νέο σύστημα. Σε σχέση με το μενού τώρα, τον κατάλογο και τις συζητήσεις που είχαμε διάφορους συναδέλφους τους τελευταίους μήνες. Και για να προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτούς τους συναδέλφους, έχοντας πλήρη επίγνωση ε, της ε, ε θα έλεγα, ε, θέσης ε, της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής για το μενού, προσπάθησα λοιπόν να εισαγάγω αυτή τη νέα έννοια της οικολογικής επιστοποίησης που ουσιαστικά εξισούται με το μενού, όμως πλαισιώνεται με κοινοτικό τρόπο. Σε αυτό το μέτρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν δεχτεί την πρόταση της οικολογικής πιστοποίησης, δίνει λύση και στο θέμα του μενού, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μενού και αποφεύγουμε έτσι τις ατέρμονες συζητήσεις, διότι αυτό που έχει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να διαπιστώσει πόσο αμφιλεγόμενα είναι τα ζητήματα της διαφοροποίησης των ε, ε, καλλιεργειών, το ζήτημα των ε, μονίμων μόνων. Υπάρχουν αυτά τα τρία ζητήματα τα οποία ε, θα ρυθμιστούν με 20 διαφορετικά μέτρα για να μπορέσει να εφαρμοστεί το σύστημα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ ανταυτού προτείνω ένα σύστημα τη οικολογική τυποποίηση, το οποίο είναι ικανό να μα δώσει τη λύση και θα ήθελα να σα υπενθυμίσω παρεπιπτόντω ότι στην περίπτωση του μενού Εάν δεν μετακινηθεί από τη θέση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα έχουμε ως αποτέλεσμα την εξάρτηση από την ομοφωνία του Συμβουλίου. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι εφικτή η ομοφωνία του Συμβουλίου για να συμπεριληφθεί το μενού στο πρασίνισμα του πρώτου πυλώνα και γι' αυτό σας λέω ότι η δική μου πρόταση είναι πιο ρεαλιστική και δράζεται σε μια πιθανή ε, συμβαστική λύση, μια εφικτή συμβαστική λύση. Ελπίζω λοιπόν με αυτή την πρόταση να υπάρξει μεγαλύτερη προσέγγιση ε, σε σχέση με την ε, ε, άκαμπτη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα για τα θέματα του κυρίου Μποβέ και του κυρίου Ντάντα, η άμυψη σπορά. Είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει επανειλημμένα στο παρελθόν. Όσοι έχουν γεωπονικές γνώσεις γνωρίζουν ότι η άμυψη σπορά είναι μια λύση για το περιβάλλον πολύ καλύτερη από την διαφοροποίηση και την εναλλαγή των καλλιεργειών διαφορά έγκυται στους μηχανισμούς ελέγχου. Για να ελέγξει κανείς ε, την έκταση με δορυφόρο, ε, αν υπάρχουν ε, μία, δύο ή τρεις καλλιέργειες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όμως, για να καταλάβουμε ποια είναι η ετήσια διαδοχή των διαφόρων καλλιεργειών μέσω δορυφόρου, κατά τη γνώμη μου και εγώ σας ξέρω, είναι κάτι το αδύνατο. Γιατί λοιπόν προτείνεται αυτή η αναλλαγή καλλιεργειών, όχι επειδή δεν συμφωνεί για την ε, για το ότι η άμυψη σπορά ε, είναι φιλική προς το περιβάλλον, αλλά διότι πρέπει να συνειδητοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να είναι εφικτός και ο έλεγχος και να είναι απλός ο έλεγχος. Ε, πρέπει να έχουμε κάποια συνοχή και ηρμό στις προτάσεις μας. Επιδιώκουμε την απλούστευση, άρα θέλουμε και απλούστερους ελέγχους και ζητούμε λοιπόν να αντικαταστήσει την αλλαγή των καλλιεργειών με την άμυψη σπορά. Θα ήθελα σε σχέση με αυτό που μα είπε η Ελίζα στην ΚΕΡΕ, να προσθέσω κάποια πράγματα. Μου ζήτησαν ε, διευκρινήσει σε σχέση με όσου διαχειρίζονται τι γεωργικέ εκμεταλλεύσει. Κοιτάξτε, όταν ε, σα μιλάω για τι ε, αναδασωμένε περιοχέ και για άλλου είδου γέε, γιατί το κάνω, διότι δεν υπάρχει απαραίτητα ένα συνεταιρισμό παραγωγών. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα από τη χώρα μου, την Πορτογαλία. Περίπου 10% του δάσου είναι κοινή χρήση ούτε δημόσια είναι αυτή η γη, ούτε ιδιωτική. Και ξέρετε ποιο αναλαμβάνει τη διαχείριση, η τοπική κοινότητα. Βάσει λοιπόν τη πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλείονται αυτοί και δεν μπορούν πλέον να διαχειρίζονται αυτέ τι γη. Δέχομαι ότι σε κάποιε συγκεκριμένε περιπτώσει μπορεί αυτό να δημιουργήσει πρόβλημα στα κράτη-μέλη, αλλά ε, νομίζω ότι με τη δική μου πρόταση ανοίγουμε το δρόμο για να έχουμε μια ευρύτατη λύση που θα ε, μα επιτρέψει να διαχειριστούμε τέτοιου είδου αναδασωμένε ε, περιοχές. Ε, απλώς θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα πιο συγκεκριμένο ορισμό. Υπάρχουν ε, ε, διάφορα άλλα ζητήματα. Ένα λεπτάκι γιατί είπε κάτι ο κύριος Νταντάν και ήθελα να το διευκρινίσω, να το βρω στις σημειώσεις μου και επανέρχομαι. Desculpa. Sim, ναι. Είναι η περίοδος κατά την οποία γίνεται χρήση της γεωργικής έκτασης. Ε, πιστεύω ότι μπορούμε να προβλέψουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ε, και ως προς την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα θα σας ε, έλεγα ότι μέσα στα περιβαλλοντικά μέτρα θα πρέπει να συμπεριλάβουμε το 30% των κονδυλίων για αυτά τα αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα καθώς και για την εφαρμογή της οδηγίας σε πλαίσιο για τα ύδατα. Ε, ε, φυσικά χρειαζόμαστε ταυτόχρονα ε, δίκαιους όρους ε, ανταγωνισμού σε σχέση τώρα με μια επανερχόμενη κριτική, δηλαδή ότι παραγνωρίζεται ο ρόλος της γυναίκας γεωργού στα επιμέρους μέτρα. Δέχομαι την, ε, το σχόλιο σας και θα καλύψω αυτό το χάσμα, το κενό συγγνώμη που υπάρχει μέσα στην έκθεσή μου. Διότι έχετε δίκιο, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το ζήτημα επίση. Ε, έχω πάρα πολλά ζητήματα σημειώσει εδώ. Βεβαίω, μην ξεχνάμε ότι θα έχουμε και αρκετού μήνε μπροστά μα ε, για να τα συζητήσουμε. Ε, και νομίζω δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Αυτό που χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα είναι να διατηρήσουμε όλη αυτή την επικοδομητική προσέγγιση όπω η σημερινή συζήτηση. Και είμαι πεπισμένο ότι θα καταλήξουμε σε μια ευρύτατη συνέντευξη στην Επιτροπή τη Γεωργία και ευρύτερο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι οι αρμοδιότητε συναπόφαση που ανατέθηκαν στο Κοινοβούλιο το επιτρέπουν να λειτουργήσει με αποτελεσματικότητα ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και του Συμβουλίου και είναι προς συμφέρον μας ε, να έχουμε την ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και θα εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να είναι κρατεή η θέση του Κοινοβουλίου θα μας επιτρέψει να είμαστε ισχυροί στις διαπραγματεύσεις και να επιτύχουμε μια καλύτερη γεωργική πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την δουλειά που έχετε κάνει και τη συζήτηση όλη αυτή που έγινε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Πρέπει να θυμάστε πως πρέπει ως ένα βαθμό η κοινωνική πολιτική να γίνει πιο περιφερειακή και να υπάρχει διαφορετικός ρόλος για το κάθε κράτος μέλος. Βεβαίως δεν θα συμφωνήσουμε στα πάντα στις Βρυξέλλες. Τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες έχουν το ρόλο τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τροπολογίες πριν τις 9 Ιουλίου το μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.